colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Είναι 9 και 10, τώρα να αρχίσουμε. Θα έρθουν και άλλοι, μην νομίζετε. Σας καλωσορίζω στην ολοήμερη σήμερα συνεδρίαση τη Εξεταστικής Επιτροπής μας, πολύ εντατική με πολλούς ειδικού. Ανακοινώσει Προέδρου, αν δεν έχουμε σχόλια, θα εγκριθεί η μερίσια διάταξη που το πέρασα έτσι γρήγορα. Ο κύριος ναι, διαδικαστικό μάλλον θα το χαρακτηρίζα, ερώτηση είναι. Ο κύριος Φερχόγεν έχει δώσει σημεία ζωής. Ξέρω ότι τον ψάχνει και ο κύριος Σούλτς. Ε, απάντησε. Αυτή τη φορά στο αίτημα του κυρίου Σούλτς πλέον. Αυτό ήταν από τις ανακοινώσεις μου και με προλάβατε. Δυστυχώς δεν έχω καλά νέα. Ε, θα συζητήσουμε ε, στους συντονιστές, θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχουμε 18 γλώσσες και όπως πάντα τα στο διαδίκτυο η συνεδρίαση και μπορείτε ηλεκτρονικά να βρείτε όλα τα έγγραφα. Σχέδιο αποφάσεων των συντονιστών 24 Μαΐου συνεδρίασαν και 9 Ιουνίου, πάρα πολύ εντατικά. Ε, είναι συνημένα στο φάκελό σας τα πρακτικά και αν δεν έχετε σχόλια θα θεωρηθούν εγκεκριμένα. Τώρα, ε, συζητούμε το δεύτερο εξάμεινο των εργασιών μας, το χρονοδιάγραμμα. Εκεί λοιπόν, στις 22 Σεπτεμβρίου μέχρι 17 ε, Οκτωβρίου είχε συμφωνηθεί ήδη και το υπόλοιπο για τις ειδικές ακροάσεις θα το συζητήσουν οι συντονιστές και μέχρι την άλλη φορά θα έχουμε το πλήρες πρόγραμμα. Όπως γνωρίζετε ε, θα ακούσουμε ε, εκπροσώπους των Ηνωμένων Πολιτειών από τις αρμόδιες αρχές έγκρισης τύπου οχημάτων, από κατασκευαστές αυτοκινήτων και τις λεπτομέρειες θα τις έχετε αργότερα εν ευθέτω χρόνο. Θα ήθελα να σε επιστήσω την προσοχή στο εξή γεγονός. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά αιτήματα για ακροάσεις και αποφασίσαμε στους συντονιστές να συμπεριλάβουμε πέντε επιπλέον μισές ημέρες συνεδριάσεις, δηλαδή στο δεύτερο εξάμεινο ε, μισές ημέρες. Το δεύτερο εξάμεινο θα ε, είναι πιο εντατικό από το πρώτο. Το φθινόπωρο θα είναι θερμό και πάρα πολύ φορτωμένο. Και παρακαλώ όλα τα μέλη να φροντίσουν να είναι διαθέσιμα τις συγκεκριμένες ημερομηνίες. Κανονίστε το πρόγραμμά σας. Έχετε τις ημερομηνίες Δευτέρα 11 Οκτωβρίου το απόγευμα, Τρίτη 11 Οκτωβρίου πρωί και απόγευμα, 7 ε, Νοεμβρίου το απόγευμα και 8 Νοεμβρίου το απόγευμα. Είναι Δευτέρα και Τρίτη τελευταίες μέρες. Επίσης, θα έχουμε και στο Στρασβούργο έκτακτες συνεδριάσεις, αν χρειαστεί να συναντήσουμε κάποιον εκτάκτος. Και μια τέτοια πρώτη συνεδρία θα είναι στις 4 Ιουλίου, την επόμενη Δευτέρα του Στρασβούργου το απόγευμα. Θα έχουμε δύο θέματα. Ε, την παρουσίαση μελέτη που εμείς αναθέσαμε σε Επιτροπή ω προς τις ε, νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις μετρήσεις καυσαερίων, εκπομπών δηλαδή, και θα ακούσουμε και τον κύριο Γιος Ντίνξ ε, από το Transport και Environment. Και έρχομαι τώρα στον κύριο Φερχόιγκεν. Όπως γνωρίζετε, επίσημα απέρριψε την ε, ε, επίσημη κατά τα άλλα δική μας πρόσκληση της Επιτροπής και δική μου. Κατόπιν αιτήματος των συντονιστών έστειλα στον κύριο Σούλτς ένα mail και του ζήτησα να παρέμβει. Όπως και έπραξε, έστειλε επιστολή, απάντηση δεν πήρε συζήτησα μαζί του και άτυπα. Δεν φαίνονται πάρα πολύ καλά τα πράγματα, για να είμαι ειλικρινής. Ας προσπαθήσουμε άλλη μια φορά. Ο κύριος Σόλτς θα έχει μια και με τον κύριο Γιούνκερ και θα επανέλθουμε σε αυτό ε, στις συζητήσεις για τα συμπεράσματά μας, αλλά πρέπει να γίνει ειλικρινή συζήτηση και να καταλάβει και ο κύριος Γιούνκερ ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής νυν ότι είναι απαράδεκτο αυτό και ανάρμοστο πρώην επίτροποι να μην έρχονται στην επιτροπή μας. Μα θα πρέπει να λογοδοτούν για πράγματα που έκαναν όταν ήταν επίτροποι. Δεν επαλλάσσονται. Α, ναι, ξέχασα να πω. Ε, δέχτηκε η απάντησή του ε, στο αίτημά μας, η απορριπτική, είναι να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα. Ωραία, είναι πάρα πολύ υπέρ της διαφάνειας. Αυτό ήταν το τελευταίο που είχα να σας πω για το συγκεκριμένο θέμα. Και μέχρι την επόμενη φορά θα πρέπει να αποφασίσουμε τι συνέχεια θα δώσουμε. Ανεξαρτήτως του γεγονός θα το θέσουμε υπόψη, του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο κ. Σούλτς ο ίδιος. Κυρία Πρόεδρε, Επιτρέψτε μου συμπληρωματική ερώτηση. Ο κ. Σούλτσε, τόσο γρήγορα που το είπατε δεν τα κατάλαβα. Σήμερα λοιπόν πώς έχει κατάσταση. Ο ε, επίτροπο, πρώην επίτροπος Φερχόγεν του Σοσιαλιστικού Γερμανικού Σοσιαλδημοκρατικού κόμματο, αρνείται. Ε, αρνήθηκε επίσημα, ε, το απάντησε και θα βάλουμε την απάντησή του στην ιστοσελίδα. Ισχυρίζεται ότι σήμερα οι υπάλληλοι τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζονται από αυτών των θεμάτων είναι σε θέση να απαντήσουν καλύτερα σε αυτά τα θέματα. Εμείς θα το φέρουμε στο υψηλότερο επίπεδο, ε, όχι μόνο το Κοινοβούλιο, τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Πρόεδρο. Απολύτω, ναι. Um, uh, Έγκριση των πρακτικών τη συνεδρίασης μα 28 Απριλίου 2016. Και αν δεν έχετε άλλα σχόλια για τις ανακοινώσεις, ε, τα πρακτικά και την ημερήσια διάταξη, ε, από ό,τι βλέπω όχι, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε στην ακρόαση. Καλωσορίζουμε την κυρία Ντοροτέ Σάρ επικεφαλής ε, του αντίστοιχου τμήματος για τις μεταφορές και την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα της Deutsche Umwelthilfe, που σημαίνει η Γερμανική Οργάνωση για την προστασία και βοήθεια στο περιβάλλον. Είναι μία ΜΚΟ, ε, συμμετέχουν διάφοροι ενδιαφερόμενοι εκεί, με διάλογο ε, και προσφεύγουν διάφοροι πολίτες ενδιαφερόμενοι που θεωρούν ότι ένα έργο απειλεί το περιβάλλον, ε, την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα κτλ. Θα σας δώσουμε το λόγο εισαγωγικά για 10 λεπτά και μετά θα ακολουθήσει η συζήτηση. Ε, το πολύ ε, μία ε, ώρα και 40 λεπτά. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε και σας ευχαριστούμε πολύ και για τις απαντήσεις σας στις γραπτές ερωτήσεις. Ήταν σαφέστατες, πάντως σίγουρα θα υπάρξουν κι. άλλες. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Yeah, Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την δυνατότητα να μιλήσω σήμερα εδώ. Θα ήθελα να πω πρώτα λίγα λόγια εισαγωγικά γιατί μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Η ρήπανση του αέρα αποτελεί σημαντική πηγή ε, ασθενειών και πρόωρων θανάτων στην Ευρώπη. Σύμφωνα με ε, την έκθεση για την ποιότητα του αέρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος ε, το 2012, 72.000 πρόωροι θάνατοι οφείλονται στην έκθεση στο διοξίδιο του αζότου. Νομίζω ότι γνωρίζετε τα στοιχεία αυτά, αλλά ήθελα να το υπογραμμίσω αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ρόλο που μα ενδιαφέρει το συγκεκριμένο θέμα. Επίση, ε, ένα εκατομμύριο ε, έτη ζωή χάνονται ε, λόγω ακριβώ αυτού του ρήπου μόνο. Και οι ανώτετε τιμέ για το διοξίδιο του αζότου στην Ευρώπη παραβιάζονται σε πολλά μέρη στην Ευρώπη, ιδιαίτερα κοντά σε δρόμους με πολλή κυκλοφορία και η βασική πηγή είναι τα αυτοκίνητα δίζελ και η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μετά την εισαγωγή των ε, αυτοκινήτων, των ΙΟΤΑΧΗ δίζελ Euro 5 και Euro 6 και γι' αυτό ε, ο οργανισμός μας ε, ασχολείται με την ευελτίωση της ποιότητας του αέρα εδώ και πολλά χρόνια. Επικεντρωνόμαστε κυρίως στην ρήπανση του αέρα στις πόλεις και στις επικίνδυνες εκπομπές από δικές μεταφορές και άλλες πηγές. Στο παρελθόν ε, έχουμε δημοσιεύσει ε, διάφορες ε, μελέτες για να τονίσουμε την ανάγκη για ανάληψη δράσης για να βελτιωθεί η ποιότητα του αέρα στην Γερμανία και στην Ευρώπη. Ζητήσαμε καλύτερη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και θα βρείτε στις γραπτές μου απαντήσεις ε, αναλυτικά τις δραστηριότητές μας. Ε, το πρόβλημα του οξυδίου του αζότου είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. και στις ε, αρμόδιες αρχές ε, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και στους επιστήμονες ε, και μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Παρόλα αυτά, Πιστεύω ότι δεν έχουμε αναρωτηθεί γιατί υπερβαίνουμε τις οριακές τιμές και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε κάτι τέτοιο. Και πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανονισμό που δίδει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές. Η Υπηρεσία Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Πολιτειών ε, επίσης ε, έχει ξεκινήσει τις έχει ξεκινήσει δραστηριότητε ε, και χρειάζεται να γίνουν δύο πράγματα. Να βρούμε καλύτερε διαδικασίε στο μέλλον και να σταματήσουμε τι εκπομπέ οξυδίων του αζότου από των ε, στόλων αυτοκινήτων που έχουμε αυτή τη στιγμή. Ποιο είναι λοιπόν ο στόχο μα. Ο στόχο μα είναι να πετύχουμε πλήρη εφαρμογή τη ισχύουσα ε, νομοθεσία ε, για την ποιότητα του αέρα, για να έχουμε καθαρό αέρα για του Ευρωπαίου πολίτε. Και αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η απόδοση των αυτοκινήτων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε την συμμόρφωση των αυτοκινήτων Euro 5 και Euro 6 και θα πρέπει να ε, εξετάσουμε τα επίπεδα ρήπανσης, τα οποία οφείλονται αφενός ε, στην πολυκυκλοφορία, αλλά και στον μεγάλο αριθμό των ανθρώπων που εκτίθενται στους ρήπους. Έχουμε λοιπόν τώρα την εισαγωγή νέου κύκλου δοκιμών WLTP, καθώς και την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, να αναθεωρηθεί το πλαίσιο για την έγκριση τύπου των αυτοκινήτων. Η μελλοντική νομοθεσία θα απαιτεί έναν καλύτερο μηχανισμό ελέγχων για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση. Αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να βρούμε μία λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δηλαδή να εξετάσουμε τον στόλο αυτοκινήτων που έχουμε αυτή τη στιγμή και τα αυτοκίνητα που θα ε, πολιθούν στο εγγύσιο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι απαραίτητο για να σώσουμε ζωές ε, και για να ε, αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη στην ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία και την ευρωπαϊκή πολιτική. Επικροτούμε την απόφαση της ε, Επιτρόπου Μπιενκόφσκα να απορρίψει την προσέγγιση του δικού μας Υπουργού Μεταφορών του κυρίου Ντόπριντ. Η υπερβολική χρήση συσκευών απάτης δεν οφείλονται στην ασαφή νομοθεσία. Πιστεύουμε ότι είναι σαφής ο κανονισμός, είναι ασθενής η εφαρμογή του. Και αυτό είναι και το αποτέλεσμα μιας ε, νομικής γνωμοδότησης της ε, επιστημονικής υπηρεσίας ε, του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Και όπως θα γνωρίζετε έχουν γίνει δοκιμές σε διάφορα μοντέλα αυτοκινήτων και το πρόβλημα με τη Volkswagen δεν είναι πρόβλημα της Volkswagen, είναι πρόβλημα με τα αυτοκίνητα diesel. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, τα συστήματα εκπομπών του Opel Zafira δεν λειτουργούν σωστά το 83% του χρόνου. Και αυτό οδηγεί σε μεγάλες εκπομπές και μόνο από αυτό το μοντέλο αυτοκινήτων. Οι αρμόδιοι από όλα τα επίπεδα θα πρέπει να φροντίσουν τα αυτοκίνητα που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα είτε να ε, τροποποιηθούν είτε να απομακρυνθούν από τους δρόμους. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την εισαγωγή σας. Ξέρετε το σύστημα συνάδελφοι. Στο πρώτο γύρο θα έχουμε δύο εισηγητές και εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων και μετά θα ακολουθήσουν έρωτα ε, απαντήσεις. Ζάλμπα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την κυρία Σάρα που είστε μαζί μας και απαντήσατε στο ερωτηματολογιό μας. Στις απαντήσεις σας στις γραπτές ερωτήσεις λέγεται ότι τον Φεβρουάριο του 2011 και επανειλημμένα ενημερώθηκε η γερμανική κυβέρνηση για μια στιγμή λέω It's okay? Yes. Thank you. για μια ακόμη φορά σας ευχαριστώ που απαντήσατε και στο ερωτηματολόγιο το γραπτό που έχει σημασία για μας. Λέτε ότι έχει αποστα... είχαν αποσταλεί επιστολές στο... στη γερμανική κυβέρνηση η οποία είχε απαντήσει ότι με τους νέους τύπους ελέγχου θα έπρεπε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Εσείς ε, τι πιστεύετε ότι έπρεπε να είχαν κάνει εκείνη τη στιγμή το 11 έτσι ώστε να αποφύγουμε αυτό το οποίο συνέβη εν το μεταξύ. 2011 and... Νομίζω ότι το 2011 αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ζητήσαμε από τις γερμανικές αρχές να ξεκινήσουν τη δική τους έρευνα. Αν είχαν αντιδράσει τότε και αν είχαν ξεκινήσει μια διερευνητική διαδικασία, αν είχαν εξετάσεις, εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι εκπομπές και τι συμβαίνει με τις λεγόμενους μηχανισμούς απόκρυψης, τότε θα βρισκόμασταν στη φάση που βρισκόμαστε σήμερα πριν μερικά χρόνια. Είχατε εντωμεταξύ ε, επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή με άλλα όργανα ή με άλλες χώρες της Ένωσης. By that time we have not... Στην φάση αυτή δεν είχαμε στραφεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Υπήρχαν κάποιες έρευνες από την Γερμανική Περιβαντολογική Υπηρεσία, οι οποίες ήταν εν γνώση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς στείλαμε πάντως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα αποτελέσματα των τεστ που είχαμε κάνει από σε ποιον είχατε στείλει τα αποτελέσματά σας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπατε ότι τους είχατε στείλει τα αποτελέσματά σας. Σε ποιον τα είχατε στείλει. Στην Επίτροπο Βιευκόσκα, στον κύριο Μπάλτς. Στον κύριο Μπέγια, αν ακούσαμε καλά. Και το τελευταίο, είχατε επίγνωση του γεγονότος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, είχε τότε στοιχεία και άρχισε να εργάζεται το 2009 ε, στα πλαίσια των πραγματικών εκπομπών έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι η πρώτη στον κόσμο που να χρησιμοποιήσει επίσημα στοιχεία για ε, συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Δηλαδή εσείς το ξέρατε αυτό ότι συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το ψάχνετε. Ναι. Είχατε γνώση αυτό του γεγονότος. Ειλικρινά εγώ προσωπικά όχι. Ήξερα ότι γινόταν μια συζήτηση για να βελτιώνονται οι συνθήκες δοκιμή στο εργαστήριο, όχι σε πραγματική οδήγηση, αλλά ε, αυτό το έμαθα μόνο για τα βαρέα οχήματα, για τα φορτηγά, ότι προσπαθούσαν να βελτιώσουν τις μετρήσεις στο δρόμο. Ευχαριστώ κύριο Γκερμπράντι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και σας κυρία Σάρ για τις πρώτες απαντήσεις και την αρχική σας τοποθέτηση. Σας καλωσορίζω στην Επιτροπή μας. Έχω πολλές τεχνικές ερωτήσεις εγώ. Τι αυτοκίνητα ψάξατε, τι ερευνήσατε, με ποια μεθοδολογία, με ποια τεχνολογικά θέματα ασχοληθήκατε, τι ψάξατε το 2007. Αλλά ε, θα μπορούσατε να μας απαντήσετε γραπτώς, αλλιώς θα χαθούμε εδώ, θα πάμε όλο τον χρόνο στα τεχνικά. Αυτό που θα ήθελα να εστιάσω είναι οι επαφές σας με τις επίσημες αρχές. Είπατε μόλις ότι δεν ενημερώσατε το 2007 τις ευρωπαϊκές αρχές, μόνο το Σεπτέμβριο του 2015. Ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να μάθω ποιες ήταν οι απαντήσεις των γερμανικών επισήμων κρατικών αρχών, οι επίσημες και οι άτυπες, αφού τους ενημερώσατε από το 2007 και μετά για τα αποτελέσματά σας. Τι σας απάντησαν εκείνοι. Η απάντηση ήταν ότι βεβαίως υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις μετρήσεις ε, που γίνονται στο εργαστήριο για την έγκριση του τύπου και ε, τις πραγματικές εκπομπές ε, στην οδήγηση στους δρόμους. Δεν μου απάντησαν αν έθεσαν ε, εκπόνηση μελέτης δική τους για το χάσμα και τη ψαλίδα που υπάρχει ε, ανάμεσα στις μετρήσεις στο δρόμο και στις μετρήσεις στο εργαστήριο που σήμερα είναι κατά μέσο όρο 40%. Ε, ούτε απάντησαν να θα λάβουν υπόψη τις υψηλές εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Εγώ ξέρω ότι χώρες σαν τη Γερμανία ε, έχουν συνήθως επίσημες επαφές με γραπτή μορφή κτλ. κτλ αλλά και άτυπες επαφές ε, μεταξύ ε, δημοσίων υπαλλήλων και ΜΚΟ. Εσείς πήρατε τίποτα άτυπες απαντήσεις, ανεπίσημες, από ανθρώπους σε χαμηλότερο επίπεδο υπαλλήλων. Σας είπε κανείς ότι έχετε απολύτως δίκιο, αλλά εμείς δεν έχουμε ακόμα επίσημη αντίδραση. Ε, έτσι αποκομίσατε την αίσθηση ότι στο Γερμανικό Υπουργείο κάπου κάποιος μπλόκαρε αυτή την υπόθεση. Άτυπα, ναι, είχα την αίσθηση ότι γνωρίζανε πολύ καλά τα προβλήματα, αλλά όπως το λέτε, άτυπα, ναι, ανεπίσημα. Ωραία, ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το στοιχείο. Θα ήθελα τώρα να εστιάσω στο μέλλον. Στις γραπτές σας απαντήσεις αναφέρεται επίσης ότι ε, το, η νέα δοκιμή ε, RDE ε, δείχνει ότι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων προσπαθούν και πάλι να εξαπατήσουν με βάση τα στοιχεία αυτά στις νέες δοκιμές. Μπορείτε λίγο να το εξηγήσετε αυτό. Έχουμε κάποιες νέες αποδείξεις. Εμείς δεν έχουμε ζητήσει από τους εμπειρογνώμονές μας να εξετάσουν σε βάθος αυτά τα περίπλοκα, τις περίπλοκες τεχνικές αποδείξεις. Πάντως υπάρχουν ενδείξεις ότι στον έλεγχο RTE on board or if you drive with your um, Sorry. <laughs> Από ε, ορισμένε συνθήκες οδήγησης, σε πάση περιπτώσει, και ιδιαίτερα με κάποιες από τις δοκιμές αυτές απαιτείται να οδηγεί κανείς με ανοιχτό το παγκάζ. Ε, αυτοί είναι κάποιοι από τους δείκτες τους οποίους έχουμε θέμα. Αυτά τα οποία είδαμε στο παρελθόν είχαν σαν στόχο να αναγνωρίζουν τον κύκλο των δοκιμών και τους κανόνες κάτω από τους οποίους διεξάγεται ο κύκλος αυτός των δοκιμών και αυτό θα πρέπει να ισχύσει και στα πλαίσια του RDE, του Real Drive Emissions, για τους ελέγχους της παραγωγή, στην παραγωγή από τις υπηρεσίες ε, εποπτείας της αγοράς. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα ούτε σε εμά εδώ. Εσείς τι θα πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει σε σχέση με αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Θα μπορούσαν να ελέγχονται τα υποκατασκευή αυτοκίνητα ή κατά τη διάρκεια τη χρήση τους Κοιτάξτε, οι ίδιοι οι κατασκευαστές ελέγχουν τα αυτοκίνητά τους και καταθέτουν τις αναφορές τους στις αρμόδιες αρχές στη Γερμανία. Και γενικά τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Έχουν υπάρξει βέβαια ορισμένες μετρήσεις από την υπηρεσία την Ομοσπονδιακή του Περιβάλλοντος στη Γερμανία και θα υπάρξουν και στο μέλλον. Αλλά για τα τελευταία χρόνια δεν υπήρξε χρηματοδότηση για τέτοιου είδους μετρήσεις. Νομίζω ότι στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε μια αρχή, μια υπηρεσία διαφορετική από την υπηρεσία έγκρισης τύπου η οποία αυτή τη στιγμή εγκρίνει και ελέγχει τα αυτοκίνητα τα οποία χρησιμοποιούνται. Δεν πρέπει να ερκεστούμε σε αυτό το οποίο ισχύει σήμερα. Υπάρχει και ένα θέμα διαφάνειας, αυτό σημαίνει δημοσίευση ε, των αποτελεσμάτων αυτών των ελέγχων. Κύριος Κάρινς, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Τα διάβασα όλα αυτά που στείλατε. Εσείς η οργάνωσή σας, ε, στις γραπτές απαντήσεις σας και συνεχίζω με μια γενική ερώτηση. Ξαναδιαβάζω αυτό τον καιρό τον κανονισμό για το άρθρο 5 εδάφιο 2 παράγραφος 2 ε, για τις συσκευές αυτές που εξαπατούν και λέει ότι θα πρέπει να απαγορεύονται. Και στην επόμενη πρόταση λέγει ότι η απαγόρευση δεν θα πρέπει να ισχύει στις εξής περιπτώσεις. Όπου είναι δικαιολογημένη η ε, χρήση και τα λοιπά για να λειτουργεί ασφαλώς το αυτοκίνητο και προναλαμβάνονται τα ε, ατυχήματα. Λοιπόν, πρώτα λέει ου ε, χρησιμοποιήσεις και μετά λέει εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται με τρόπο πάρα πολύ ασαφή. Και έχουμε και αυτό το σύστημα ε, ελέγχου του τύπου και έγκρισης που δεν είναι ένα αυτοκίνητο που πάει και το ελέγχουν και περνάει, αλλά εκατομμύρια πράγματα, λεπτομέρειες που ελέγχονται σε διαφορετικά σημεία. Δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός έλεγχος. Και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι μάλλον του παρατηρητή παρά του συμμετέχοντα. Και δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι γίνεται και με τη χρηματοδότηση αυτών των εργαστηρίων, ε, των ε, συνεργείων που τα ελέγχουν, χρηματοδοτούνται από την αυτοκινητοβιομηχανία και πώς. Όλο αυτό το σύστημα δηλαδή κάπου συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα. Θα συμφωνούσατε κι εσείς με αυτή την εκτίμηση. Είναι έτσι συστημική η ε, ζημιά σε όλα τα επίπεδα, αρχής γενομένης από την νομοθεσία μέχρι ε, τις μάλλον ατυχείς διαδικασίες εφαρμογής του νόμου. Τι θα λέγατε γι' αυτό. Δεν θα συμφωνούσα Νομίζω ότι θα πρέπει να διαβάζει κανείς τον κανονισμό από την αρχή, από τις αιτιολογικές σκέψεις που λέει ότι ε, ο κανονισμός αυτός ε, στόχο έχει να συμβάλλει στην καλύτερη ποιότητα του αέρα και έτσι έχουν τεθεί τα πρότυπα. Υπάρχουν αρκετές παράγραφοι που αναφέρονται στη συμμόρφωση με τα πρότυπα εκπομπών. Σε μία συγκεκριμένη παράγραφο λέει ότι η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για να μειώσει τις εκπομπές θα πρέπει να λειτουργεί υπό κανονικές συνθήκες, υπό τις συνθήκες που βρίσκει κανείς στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι αυτό το in normal use υπό κανονικές συνθήκες είναι πολύ σημαντικό. Το ίδιο ισχύει για τα φρένα, για βαλβίδες ασφαλείας, για χιλιάδες στοιχεία ασφαλείας του αυτοκίνητου και κανείς δεν θα συμφωνούσε ένα φρένο ή μια βαλβίδα ασφαλείας ε, να λειτουργεί μόνο εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 22 βαθμούς. Αυτή λοιπόν η ρήτρα που αναφέρατε στο άρθρο 5, η ρήτρα παρέκκλησης, θα πρέπει να θεωρηθεί παρέκκληση και ε, θα πρέπει να εφαρμόζεται για την αποφυγή ατυχημάτων. Αλλά σας έδωσα το παράδειγμα του Opel Zafira που δεν λειτουργεί σωστά. Ε, πάνω από το 80% του χρόνου και τα χαρακτηριστικά που βρήκαμε στο Zafira δηλαδή το σύστημα να κλείνει όταν ξεπερνάει κανείς ε, τα 145 χιλιόμετρα την ώρα ή όταν ε, οι στροφές του κινητήρα ξεπερνούν ένα συγκεκριμένο αριθμό. Αυτό το θέμα δεν συνδέεται με κάτι τεχνικό. Ναι, συμφωνώ με αυτό που λέτε, αλλά η δυσκολία που βλέπω εγώ είναι ότι μπορεί κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ ή κατά του κανονισμού. Εσείς ε, διαβάζετε κάποια κομμάτια, τα ερμηνεύετε με κάποιο τρόπο, αλλά διαδικασία ελέγχου που έχουμε για την εφαρμογή τη οδηγία υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει μια κεντρική αρχή που να μπορεί να κάνει ανεξάρτητους ελέγχους. Και αυτή τη δυσκολία βλέπω εγώ. Έχουμε τον νόμο από τη μία πλευρά, αλλά έχουμε έναν πολύ ελλειπή μηχανισμό. Ακόμα και αν θεωρήσει κανείς ότι ο νόμος είναι απόλυτα σαφής, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι, αλλά είναι πολύ ασθενής ο μηχανισμός που υποτίθεται ότι πρέπει να διασφαλίσει την εφαρμογή του νόμου. Ε, έχουμε μία ε, πολύ διαφοροποιημένη, σκορπισμένη προσέγγιση όσον αφορά την έγκριση τύπου. Η κυρία Σάρ. Καμία νομοθεσία δεν απαγορεύει την ε, γερμανική αρχή για την έγκριση τύπου να διεξάγει μόνη της, ε, τους ελέγχους. Ή να αναρωτηθεί γιατί συμβαίνουν όλα αυτά στις Ηνωμένε Πολιτείες χρησιμοποιούνται τρόποι να υποβάλλονται αναλυτικές ερωτήσεις προς τους ε, κατασκευαστές αυτοκινήτων. Μπορεί λοιπόν ε, να ε, επικαλεστεί κανείς το άρθρο 5 παράγραφος 2. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σδάνς. Σας ευχαριστώ κυρία Σάρ που βρίσκεστε εδώ σήμερα και σας ευχαριστώ και για τις γραπτές σας παρατηρήσεις ε, που ήταν πολύ χρήσιμες στην έρευνά μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις ε, διατάξεις αναστολής ε, και τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Είδαμε αποτέλεσμα, τα αποτελέσματα δοκιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη Γερμανία. Στη Γερμανία 48 αυτοκίνητα από τα 53 έδειξαν πολύ υψηλότερε ε, εκπομπές ε, όταν ε, ξεκινούσαν με κρύο κινητήρα σε αντίθεση με αν ξεκινούσαν με ζεστό κινητήρα. Και βέβαια αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ενδεικτικό της χρήσης μιας ε, ε, συσκευή απάτης, ε, συστήματος αναστολής στα οχήματα αυτά ή πιστεύετε ότι μπορεί να οφείλεται αλλού. Η κυρία Σάρ, δεν έχω κάποια τεχνική εξήγηση γι' αυτό. Οι εκπομπές θα έπρεπε να είναι χαμηλότερες όταν ξεκινάει ο κινητήρας και είναι ήδη θερμός. Ο κύριος Τάνς. Γνωρίζουμε τι έκανε το λογισμικό της Volkswagen, διότι το ανακαλύψαμε προφανώς. Αλλά υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου υπάρχει μια συσκευή που διαχέει στο εξωτερικό μια υψηλότερη θερμοκρασία. Ή διαπιστώσαμε να τίθεται σε λειτουργία ένας μηχανισμός ε, σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Πιστεύετε ότι οι κατασκευαστές έχουν βάλει στο λογισμικό μια σειρά τέτοιων ορίων και να είναι πολύ πιο ευρεία η χρήση συστημάτων αναστολής ε, υπό διαφορετικές μορφές ε, και ακολουθώντας διάφορες ερμηνείες του ε, ισχύοντος κανονισμού. Αν πάρουμε το παράδειγμα των 100... Αν πάρουμε το παράδειγμα των 145 χιλιόμετρων ε, την ώρα, αυτό σίγουρα ε, είναι εκτός ε, των ορίων του επίσημου κύκλου ελέγχων, όπως και το όριο στροφών του κινητήρα. Η θερμοκρασία εντός του εργαστηρίου είναι 20 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να Ξανααναφέρω λοιπόν το Opel Zafira που δεν θέλω να το κατηγορήσω στο μόνο κακό αυτοκίνητο εδώ μέσα αλλά η Opel λέει ότι το σύστημα μείωση των εκπομπών λειτουργεί τέλεια σε θερμοκρασία 20 με 30 βαθμούς Κελσίου. Και υπάρχει συζήτηση εάν κλείνει η συσκευή μετά από 22 λεπτά, διότι ο κύκλος δοκιμών διαρκεί 20 λεπτά. Τι να σας πω. Μάλλον έχετε δίκιο. Ωραία. Λοιπόν, για τα συμπεράσματά σας τα παρατηρήσαμε. Κάτι το οποίο προσπαθούμε εδώ να δούμε. Και μετά από τα αποτελέσματα, τα παραδείγματα που δείχνουν για τις συσκευές παραπλάνησης και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπέμπουν τα αυτοκίνητα ή μας λένε ότι εκπέμπουν, στην αρχή για τα ε, επαγγελματικά οχήματα και αργότερα και για τα υπόλοιπα οχήματα με τα οποία ασχολείται και η δική σας οργάνωση τα τελευταία δέκα χρόνια. Ποια ήταν χοντρικά η αντίδραση στα ευρήματά σας, στα συμπεράσματά σας και στις προτάσεις σας. Οι αντιδράσεις των αρχών ήσαν επαρκείς, Πιστεύετε ότι ελήφθησαν εγκαίρως υπόψη με κατάλληλο τρόπο και ποιος το έκανε ή δεν το έκανε αυτό. Νομίζω ότι οι αντιδράσεις της δημοσιεύση μας και στα, στα αιτήματά μας ήταν ανεπαρκείς. Και δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν αν το EPA δεν είχε δημοσιεύσει αυτά τα οποία δημοσίευσε με τον τρόπο που τα δημοσίευσε. για τη γερμανική αρμόδια αρχή υπήρξε διστακτική αντιμετώπιση για την αντιμετώπιση των ευθυνών στην αυτοκίνητο βιομηχανία και για να υπάρξει πλήρη συμμόρφωση της νομοθεσίας στη νομοθεσία. Ο επόμενος κύριος Χένκελ. Προτιμούσα να μιλήσω γερμανικά. Καταλαβαίνετε γερμανικά, έτσι δεν είναι. Στην ε, απάντησή σας αναφέρετε ότι σε κάποιες δοκιμές ε, έχει ληφθεί υλικό από την Toyota. Ρωτώ λοιπόν, έχετε προσπαθήσει να λάβετε υλικό και από άλλες εταιρείες και το υλικό που χρησιμοποιήσατε, ε, πώς θα το βαθμολογούσατε όσον αφορά την αξία του υλικού. Τι ακριβώς ε, εννοείται. Ο κύριος Χένκελ γράφει εδώ. Γράφεται ότι τα φίλτρα αυτά αναφέρθηκαν από την Toyota ως παράδειγμα. Στη σελίδα 4 της γραπτής σας απάντησης αναφέρεται αυτό. Έχετε λάβει λοιπόν υποστήριξη όσον αφορά την αξιολόγηση της μείωσης ε, των εκπομπών από την Toyota. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, έχετε λάβει αντίστοιχη υποστήριξη από άλλη εταιρεία, μπορείτε να μου απαιτήσετε στα γερμανικά. Η οικονομική υποστήριξη από πλευρά της Toyota ε, πραγματοποιείται εδώ και 15 χρόνια πενταψήφια ποσά για πενταψήφια ποσά πρόκειται και κάθε χρόνο υποβάλλουμε σχετικά αιτήματα στα Υπουργεία, στις επιχειρήσεις του DAX 100. για να ε, δούμε σε τι βαθμό ε, ε, υπάρχει αυτή η συνείδηση για το περιβάλλον και όσον αφορά τα αυτοκίνητά τους. Και από άλλες εταιρείε από τον Σεπτέμβριο του 2010 δεν έχουμε λάβει σχετική βοήθεια. Επόμενη ερώτηση. Προηγουμένως είπατε και εξεπλάγει λίγο ότι δεν είναι σκάνδαλο Volkswagen αυτό, αλλά είναι σκάνδαλο των πετρελοκινήτων αυτοκινήτων. Καλά, δεν θα πρέπει να γίνει και εκεί μια διάκριση αυτά που έκανε η Volkswagen με τη συσκευή εξαπάτησης, το defeat device και ε, με αυτή τη δήλωσή σας μπορεί να προκληθεί εντύπωση ότι εξαπατούν όλοι οι κατασκευαστές αυτοκινήτων Γερμανοί και άλλες αυτοκινητομηχανίες. Μα υπάρχουν διάφοροι κατασκευαστέ που στο μεταξύ το έχουν ομολογήσει ότι έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιε συσκευέ. Προσπάθησα να περιγράψω προηγουμένω ότι υπάρχουν δείκτες και κριτήρια σύμφωνα με τα οποία αντιδρούν αυτές οι συσκευέ ω προ την ταχύτητα κτλ που ε, αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει κάποια σχέση. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι να πω το εξή. Οι υψηλέ εκπομπές ε, διοξιδίου ή οξυδίων του αζότου σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης δεν είναι κάτι που προκαλείται μόνο από τα, Volkswagen αλλά από όλα τα diesel. Δηλαδή, ο κύριος Χένκελ. Ναι, καλά, αυτό το έχουμε καταλάβει και εμείς ε, μέχρι τώρα ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα ε, ότι άλλες τιμές δίνουν στο εργαστήριο οι δοκιμές και άλλες στον πραγματικό κόσμο. Αλλά θα μας βοηθούσε και εάν εσείς στην επικοινωνία σας κάνατε διάκριση ανάμεσα σε αυτή την απάτη κανονικά της Volkswagen και των άλλων διαφορετικών μετρήσεων. Δεν θα θεωρείτε σκόπιμο να το λέτε και εσείς στις ανακοινώσεις σας. Στις δικές μας ανακοινώσεις τι λέμε. Ότι τα αποτελέσματα που πήραμε από άλλους κατασκευαστές ή που τα έχουμε ψάξει ή εμείς ή άλλες οργανώσεις είναι επίσης παράνομα. Ε, είτε ε, το έχουν ομολογήσει όπως η Volkswagen είτε όχι, όπως άλλες εταιρείες που δεν, δεν ε, έχει αποδειχθεί ότι είναι σύνομες αυτές οι δράσεις. Τελευταία ερώτηση. Μιλήσατε και θα επανέλθω στο Πασάτ το 2011 και είπατε ότι το Υπουργείο δήλωσε ότι γνώριζε αυτό το πρόβλημα ότι σπαθέμετη και παράνομη πρακτική. Έχετε εσείς αποδείξεις για αυτό το πράγμα που ισχυρίζετε, μπορείτε να τις προσκομίσετε. Και διαπιστώνετε ότι το Υπουργείο πραγματικά είπε τέτοιο πράγμα. Ότι πρόκειται για παράνομη πρακτική, δηλαδή το, το παραδέχτηκε και το Υπουργείο. Έχουμε τα πρακτικά της συνομιλίας αυτής της συνεδρίασης και με τα στοιχεία που είχαμε φέρει τότε, ε, ε, καταδείξαμε το πρόβλημα ότι είναι υψηλές εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου και ότι πρόκειται για παράνομες πρακτικές. Οπότε απάντησε τότε το, Υπουργείο ότι γνωρίζει το πρόβλημα. Τώρα, αν σημαίνει ότι και το Υπουργείο τότε θεωρούσε και το κατέτασε αυτό ως παράνομο, αυτό ελέγχεται. Υπήρξε μια ερώτηση της Γερμανικής Βουλής εάν υπάρχουν στοιχεία από αυτή τη συνάντηση, πρακτικά δηλαδή των συζητήσεων, ε, στο πρωτόκολλο του Υπουργείου. Δυστυχώς δεν το έχουν πρωτοκολλήσει αυτοί. Ευχαριστώ πολύ κύριο Φέντερλε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Βεβαίως σας καλέσαμε γιατί συμφωνήσαμε στην Επιτροπή ότι εκπροσωπείται μια οργάνωση η οποία είναι και αξιόπιστη και ικανή και σχετική με τη δική μας έρευνα. Αλλιώς δεν θα σας καλούσαμε εδώ. Θα ήθελα καταρχάς να διευκρινίσω κάτι. Γίνεται μια συζήτηση σήμερα το πρωί σχετικά με την νομοθεσία, αν είναι σαφής ή όχι. Και προφανώς εδώ οι απόψεις είναι ε, σε αριθμό όσα και τα μέλη παρόντα. Αλλά από τις δικές σας γνώσεις και εμπειρία μπορείτε να πείτε εσείς ότι είναι σαφή η νομοθεσία. Ναι, εγώ θα το έλεγα αυτό, είναι σαφή η νομοθεσία. απαιτεί να χρησιμοποιείται η κατάλληλη τεχνολογία ε, ε, στις εξατμίσεις ε, των αυτοκινήτων έτσι ώστε να γίνονται σωστά οι εκπομπές. Σας είπα, για 140 χιλιόμετρα ταχύτητα, αυτό είναι μια συνήθιση ταχύτητα. Ευχαριστώ, σαφής απάντηση. Επίσης, λέτε ότι υπάρχει κάποια προθυμία από πλευράς γερμανικών αρχών να αναλάβουν κάποια δράση μετά τη δημοσίευση, ότι υπήρξε τουλάχιστον ε, των στοιχείων και μάθαμε από τις τελευταίες ακροάσεις ότι από το 2004 αναφέρεται ότι υπάρχει διαφορά στις μετρήσεις αν αυτές γίνονται στο εργαστήριο ή στο δρόμο. Άρα, εσείς λέτε ότι είναι εντάξει η νομοθεσία, αλλά το πρόβλημα πιστεύετε ότι είναι η εφαρμογή της, η παρακολούθηση και ο έλεγχος. Και ποιε θα ήταν οι δικές σας συστάσεις προς εμάς ε, που ασχολούμαστε με τη μελλοντική νομοθεσία. Τι πρέπει να κάνουμε, να οργανώσουμε ένα σύστημα Εφόσον υπάρχουν αναφορές που καταγγέλουν ότι δεν ισχύουν ε, αυτά που λέει η νομοθεσία και δεν εφαρμόζονται στην πράξη, από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα πολιτικό σύστημα, μια πολιτική μηχανή και ένα νομικό πλαίσιο που θα πρέπει να κινητοποιείται. Κάποιες ε, απαντήσεις έχουν ήδη ξεκινήσει να δίδονται. Από το 2017 θα έχουμε τους νέους ελέγχους RDE, Real Drive Emissions. Θα υπάρξει ένας νέος κύκλος δοκιμών επίσης και νομίζω ότι τα δύο αυτά μέσα θα μικρύνουν την απόσταση ανάμεσα στα αποτελέσματα των τεστ και στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι οι ανεξάρτητες μετρήσεις θα πρέπει να καταστούν τμήμα της διαδικασίας έγκρισης τύπου. Και θα πρέπει επίσης να ισχύσουν και για, να γίνουν και για τον υπάρχοντα στόλο αυτοκινήτων. Ακόμα και αν συμφωνούμε ότι υπάρχει ε, ε, μια διαφορά ανάμεσα στις εργαστηριακές συνθήκες και στις πραγματικές συνθήκες οδήγησης, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα ξεκαθαρίζεται ότι τα όρια εκπομπών τα οποία ορίζονται με τον παρόντα κανονισμό ε, δεν θα πρέπει να εκπληρούνται δεν είναι θέμα αριθμητικό, είναι μια αναγκαιότητα η βελτίωση του αέρα που εισπνέουμε. Και η τελική μου ερώτηση. Θα επαναλάβω το θέμα της νομοθετικής ρύθμισης, αν και οι απαντήσεις σας ήταν πλήρης. Καμία από τις χώρες μέλη δεν έχει ζητήσει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις τα τελευταία δέκα χρόνια, οπότε αυτό κάτι σημαίνει για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών. Στην γραπτή σας απάντηση στην ερώτηση 10, λέτε ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους έτσι ώστε να αποφύγουμε τα βρώμικα αυτοκίνητα σε εισαγωγικά, κάτι το οποίο δεν γίνεται σήμερα. Υπάρχουν πιστεύετε και άλλοι τρόποι για να παραπλανήσει κανείς τους καταναλωτές, να ε, μην εφαρμόσει τους κανόνες. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι για την ε, εξαπάτηση σε σχέση με το πραγματικό επίπεδο εκπομπών. Πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες ε, μετρήσεις. Το RDE είναι και διαδικαστική πρόταση και μέσο για την πραγματοποίηση ξεκαθαρίζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να διεξάγονται. Θα ήταν καλό να υπάρξουν συμπληρωματικοί έλεγχοι με την ίδια τεχνολογία μέτρησης που έχουμε σήμερα, αλλά κάτω από συνθήκες οι οποίες δεν θα είναι εκ των προτέρων γνωστές. Αυτό γίνεται στη ΣΥΠΑ. Ernst. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ για τα σαφή σας σχόλια. Ας αρχίσω από το θέμα ποιος ήξερε τι και γιατί αισιόπισαν οι πάντες. Από αυτά που μας λέτε κατάλαβα ότι ήδη από το 2007 ε, αντιδράσατε με συνέντευξη τύπου. Το 2009 στη συνέχεια απευθυνθήκατε στον κύριο Τίφενζε, Υπουργό Μεταφορών τότε, το 2010 στο Ραμζάουερ, Αλτμάγερ, σε διαδοχικούς υπουργούς μεταφορών, εσείς κάνατε κρούσεις. με επιστολές, με αναβολές επισκέψεων. Δεν είχαν χρόνο υπουργοί, σας παραπέμπανε σε γενικούς γραμματείς. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, πώς το εξηγείτε και Είχατε και άλλες ε, προσπάθειες και απόπειρες να συναντηθείτε με το Υπουργείο πριν ε, γνωστοποιηθεί το σκάνδαλο, πριν ξεσπάσει. Και επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το 2011 λέτε, χτυπήσατε την πόρτα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είπατε σε ποιους επιτρόπους ε, γράψατε και δεν θυμάμαι και ποιους άλλους υπαλλήλους. Καμία αντίδραση υπήρξε. Είχατε απάντηση ε, τι συνέχεια δόθηκε. Ποιος έκανε τι. Κινήθηκε τίποτα. Για να αρχίσω από το δεύτερο. Το 2011 ακόμα δεν είχαμε στείλει τίποτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τότε αρχίσαμε. Ενημερώσαμε τους τρεις επιτρόπους από το Σεπτέμβριο του 2015 με τις μετρήσεις μας. Πήραμε αριθμό πρωτοκόλλου ότι το έλαβαν ε, και ότι ευχαριστούμε πολύ και θα το παρακολουθήσουμε. Μια αυτόματη απάντηση. Μετά ε, είχαμε συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή της για το πλαίσιο για την έγκριση τύπου. Εκεί έχουμε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο παρελθόν που είχαμε επευθυνθεί στους διάφορους υπουργού, τον εκάστοτε υπουργό μεταφορών, του αναφέρατε και ονομαστικά, υπήρξαν συνομιλίε ε, σε επίπεδο τμήματα αρχών, ε, διευθυντών, κατώτερο του Γενικού Γραμματέα από το 2011 και από το Σεπτέμβριο 2015 εκ τότε δεν έχουμε επαφές με το Υπουργείο Μεταφορών. Του στείλαμε ε, τις μετρήσεις μας ε, τους ε, προσφέραμε ε, τη δυνατότητα να κάνουμε συναντήσεις, ζητήσαμε απάντηση και από τον Υπουργό και από τον Υφυπουργό και από τον Γενικό Γραμματέα, αλλά τίποτα μέχρι τώρα. Και πώς το αιτιολογούν, λέει η κυρία Έρνστ. Δεν κατάλαβαν ότι υπήρχε ανάγκη. Όχι, δεν το αιτιολόγησαν, ούτε δικαιολογήθηκαν, απλώς δεν μας απήντησαν. Ωραία. Και ένα δεύτερο τώρα να ρωτήσω, λέει κυρία Ένστ, για τις ε, συσκευές αυτές ε, ε, που ε, σταματούν τη λειτουργία. Υπάρχουν παράνομες και νόμιμες και για τον κανονισμό του 2007, είναι ο κανονισμός 750. Είπατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει ε, διαδικασίες ε, για αντίδραση και απάντηση σε παραβάσεις και παραβιάσεις. Νομίζετε ότι είναι σκόπιμο κάτι τέτοιο, πρέπει να νομοθετηθεί, πρέπει να αλλάξει κάτι ή μήπως όχι. Να ξεκινήσω από το τέλος. Δεν είμαι βέβαιη αν έχει η Κομισιόν διαδικασίες για να χειριστεί τέτοιες ε, παραβάσεις. Στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο, θα πρέπει η Κομισιόν να φροντίσει μια Ευρωπαϊκή Αρχή να ελέγχει τις ε, εθνικές αρχές ε, καθώς και να οργανώνει τους ελέγχους. Η Κομισιόν γνωρίζει ότι τουλάχιστον στη Γερμανία και οι εκπομπές ε, οξυδίων ε, του αζότου που υπάρχουν στην ε, Γερμανία ξεπερνούν τα όρια στην εθνική νομοθεσία, καθώς και η ποιότητα του αέρα δεν συμμορφώνεται με την οδηγία και γι' αυτό υπάρχει μια διαδικασία επιπαραβάση κατά της Γερμανίας. Θα μπορούσε κανείς να αναρωτηθεί πώς μπορούμε να εξηγήσουμε, να υπερβαίνουμε συνέχεια τις ε, τιμές ε, τη στιγμή που έχουμε τόσα αυτοκίνητα δίζελ στους δρόμους. Ε, έγινε αναφορά στα αυτοκίνητα Euro 5 και Euro 6 που δεν ε, συμμορφώνονταν, ε, αλλά η Κομισιόν δεν έκανε το επόμενο βήμα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Χάρμς. Καλημέρα, κυρία Ζάρ. Και εμείς σας ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνετε για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη και στις πόλεις μας. Θα ήθελα να επανέλθω στην ε, συνομιλία που είχατε τον Φεβρουάριο 2011 με το ε, αρμόδιο Υπουργείο της ε, Γερμανίας σχετικά με τις τιμές οξυδίων του αζότου. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, εκείνη ήταν η πρώτη ευκαιρία να αναφερθεί το παράνομο λογισμικό. Στην Επιτροπή μας, ε, είχαμε επίσκεψη του εμπειρογνώμονα από το Κοινό Κέντρο Ενεργών, ε, ε Ερευνών, συγγνώμη, ο οποίος ε, μας είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να θεωρήσει κανείς ότι γινόταν χρήση των διατάξεων αναστολής παρότι υπήρχε υπέρβαση των ορίων. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, εσείς πώς καταλάβατε ότι χρησιμοποιείτε το παράνομο λογισμικό. Επίσης θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν υπήρχαν άλλες τεχνικές εξηγήσεις για τις αποκλήσεις στις τιμές. Έχουμε πολλές ανταλλαγές με βιρογνώμονες από την βιομηχανία, από τον τεχνικό κόσμο, να το πω έτσι, και ανεπίσημα λαμβάνουμε διάφορες πληροφορίες. Και από ανεπίσημες ε, πληροφορίες ε, είχαμε ενημερωθεί για την ε, χρήση παράνομου λογισμικού. Είναι απαραίτητο λοιπόν κάποιος που έχει την τεχνογνωσία που μπορεί να διαβάσει το λογισμικό αυτό να βρει τον ε, τεχνικό συσχετισμό. Θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται τέτοιο λογισμικό το οποίο ενημερώνει το αυτοκίνητο ότι τώρα γίνεται δοκιμή ε, και έτσι βελτιστοποιούνται οι τιμές όσον αφορά τις εκπομπές όσον αφορά τις υψηλές εκπομπές ε, οξυδίων του αζότου. Δεν έχουμε άλλη τεχνική εξήγηση. Δεν γίνεται σωστά το φιλτράρισμα των εκπομπών. Και θα πρέπει να βρεθεί τρόπος ώστε να τηρούνται οι τιμές ε, στα ε, αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στο δρόμο και μάλιστα ε, να τηρούνται όχι μόνο οι ευρωπαϊκές τιμές αλλά και οι αμερικανικές. Ήταν λοιπόν δεν καταλάβαμε λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η υπέρβαση με τις τεχνικές γνώσεις που είχαμε. Η κυρία Χάρμς, μετά από την ε, συζήτηση αυτή στο Υπουργείο Μεταφορών τον Φεβρουάριο του 2011, δεν έχω καταλάβει ε, αν το Υπουργείο δήλωσε ότι το Υπουργείο καταλαβαίνει ότι ε, γίνεται χειραγώγηση των αποτελεσμάτων Μπορείτε να το πείτε πιο καθαρά. Υπήρξε σαφή σε δήλωση από πλευρά του Υπουργείου ότι γνωρίζουν ότι χρησιμοποιούνται διατάξει αναστολή. Και όταν ξεκίνησε η συζήτηση για τις παράνομες πρακτικές της βιομηχανίας αυτοκινήτου, υπήρξαν αιτήματα προς το Υπουργείο Μεταφορών και από ποιους, τι αιτήματα ήταν αυτά και τι βήματα έγιναν. Στην ε, συζήτηση αυτή εμείς ε, επισημάναμε ότι υπάρχουν αποκλήσεις ε, σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτων και ότι θεωρούμε ότι χρησιμοποιείται σύστημα αναστολής το οποίο κατά τη γνώμη μας είναι επίσης παράνομο. το Υπουργείο τότε είπε ότι γνωρίζει ότι υπάρχουν οι αποκλήσεις στις τιμές. Δεν θα έλεγα ότι το Υπουργείο θα μας έλεγε ότι γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούνται παράνομες ε, συσκευές αναστολής. Εμείς είχαμε πει τότε ότι η δική μας εκτίμηση είναι ότι χρησιμοποιούνται παράνομες διατάξεις αναστολής. Τότε είχαμε επανειλημμένα ζητήσει από το Υπουργείο να κάνει δικούς τους ελέγχους, να βρει τις αιτίες Και αυτό το κάναμε και με τις δοκιμές που δημοσιεύσαμε από το 2015 και μετά. Επανειλημμένα ζητήσαμε από το Υπουργείο να εξετάσει περαιτέρω τα αυτοκίνητα αυτά, διότι εμείς γνωρίζαμε ότι ανα πάσα στιγμή ελέγχουμε ένα αυτοκίνητο μόνο από κάθε ε, μοντέλο. Πρόκειται δηλαδή για δειγματοληπτικό ε, έλεγχο. Για να έχουμε λοιπόν επιπλέον στοιχεία είναι απαραίτητο οι αρχές να ξεκινήσουν δικούς τους ελέγχους. Το Υπουργείο έκανε μετρήσεις, ε, αλλά δεν ε, έχει δημοσιεύσει όλα τα στοιχεία. Για παράδειγμα, όχι τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Ε, ούτε είναι πάντα εύκολο να καταλάβει κανείς πώς έχουν καταλήξει τη συγκεκριμένη αξιολόγηση. Ευχαριστώ. Sì, grazie mille per σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψή σας, για τις απαντήσεις σας και για την πολύ χρήσιμη εργασία της οργάνωσης την οποία εκπροσωπείτε. Για την μυστικότητα τώρα, την εμπιστευτικότητα των δεδομένων των δοκιμών που έγιναν από τις διάφορες υπηρεσίες με απογοητεύει το γεγονός ότι δεν δημοσιεύονται και δεν υπάρχει διαφάνεια έτσι ώστε να γνωρίζει κανείς α, ακριβώς το τι συμβαίνει. γύρω από τις εκπομπές. Ανησυχώ από την Ιταλία δεν έχει ακόμα ε, κάνει μια πραγματική έρευνα ή αν έχει κάνει δεν έχει δημοσιεύσει τα αποτελέσματά της. Θα ήθελα να μου πείτε αν είναι δυνατόν. αν επί τη βάση των εμπειρογνωμόνων και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα μπορούμε να πούμε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα και τα κράτη-μέλη σε όλα τα επίπεδα γνώριζαν για τις διαφορές ε, των αποτελεσμάτων ανάμεσα στις εκπομπές σε περιβάλλον εργαστηριακό και σε περιβάλλον πραγματικό. Σύμφωνα με την δική σας άποψη και υπό το φως των υπαρχουσών τεχνολογιών, η καθυστέρηση με την οποία παρουσιάστηκε η πρόταση αναθεώρησης της διαδικασίας ελέγχου του νέου λεγόμενου ευρωπαϊκού κύκλου είναι κάτι το οποίο δικαιολογείται. Θα πρέπει να ξαναρωτήσω, ε, τι καθυστέρηση δημοσίευσης υπήρξε? Now Έλεγα ότι υπήρξαν κάποιες ε, γενικές σκέψεις σύμφωνα με τις οποίες η Ιταλία ακόμα δεν έχει κάνει κάποια έρευνα και δεν έχει δημοσιεύσει οποιαδήποτε έκθεση σε σχέση με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία κτλ. Ε, αναφέρθηκα στη δυσκολία που υπάρχει να δημοσιεύονται τα δεδομένα. Αλλά ε, η ερώτηση αφορά το νέο κύκλο δοκιμών. Οι αλλαγές και οι προτάσεις αλλαγών των δοκιμών, των διαδικασιών ε, ήρθε με καθυστέρηση από ό,τι φαίνεται. Προφανώς τα ευρωπαϊκά όργανα και οι εθνικές αρχές δεν έβλεπαν τη διαφορά στα, στις δύο κατηγορίες των τεστ. Να το πω στα γερμανικά. Ο νέος κύκλος δοκιμών συνδέεται στενά με την, ε, σύγκριση, με την ε, μετατροπή μάλλον των παλιών στοιχείων ε, στο, ώστε να είναι συγκρίσιμα με τα νέα στοιχεία. Και εμείς πιστεύουμε ότι έχει καθυστερήσει η διαδικασία αυτή. Διότι το επόμενο βήμα ε, για το διοξίδιο του άνθρακα, τώρα που ε, έχουν γίνει Τώρα που έχουν θεσπιστεί τα όρια για το 2020, το επόμενο βήμα είναι να θεσπιστούν και το 2025 αλλά θα πρέπει να συμφωνηθεί αυτός ο νέος κύκλος δοκιμών. Ωραία, ευχαριστώ, αλλά θα ήθελα να μου πείτε, το 2005 ήταν ήδη σαφές ότι υπήρχε άλλη μέθοδος πολύ πιο ακριβής από ε, τον ε, Ευρωπαϊκό Κύκλο Δοκιμών, ε, όπως ο κύκλος Άρτεμις. Γιατί πιστεύετε ότι επιλέχθηκε ο νέος ευρωπαϊκός κύκλος οδήγησης. Εάν είχαμε υιοθετήσει τη μέθοδο Άρτεμις, θα μπορούσε να έχει μειωθεί το χάσμα ανάμεσα στις μετρήσεις ε, υπό πραγματικές συνθήκες ε, και τις ε, μετρήσεις στο εργαστήριο. Η κυρία Σάρ, νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να κλείσουμε το χάσμα ανάμεσα στα αποτελέσματα από το εργαστήριο και τα αποτελέσματα σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης είναι να γίνει έλεγχος των αυτοκινήτων που αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν στον δρόμο. Αποφασιστικό δεν είναι το τι ε, ε, δοκιμή χρησιμοποιούμε στο εργαστήριο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο. Ε, ήμουν αρκετά επίκης με τις παρεμβάσει στον πρώτο γύρο. Ε, δεν θα είμαι τόσο επίκη στο μέλλον. Ο κύριος Γκίζεκε. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Σάρφ, ευχαριστώ που μα ήρθατε. Λοιπόν, τι μας είπατε, ότι είναι καλοί οι νόμοι, σπάνια μας επενούν για την νομοθεσία, το πρόβλημα είναι στην εφαρμογή. Εγώ δεν θέλω να διαπληκτιστώ ούτε με τον συνάδελφο Χένκελ, αν είναι ε, περίπτωση Volkswagen ή άλλων, φαίνεται ότι ενέχονται και άλλοι κατασκευαστές, ε, άλλος με λογισμικό, άλλος με συσκευή εξαπάτησης. Αυτά θα τα αποφασίσουν τελικά τα δικαστήρια, ποιος έχει παραβεί το νόμο και ποιος όχι. Εγώ θα ήθελα τώρα να στραφώ στο μέλλον, έτσι, με αισιοδοξία γιατί εμεί είμαστε μια εξεταστική επιτροπή που πρέπει να εκπονήσει συστάσει. Τώρα πέτοινος πρόκειται. Για τα πραγματικά καύσα αέρια θα πρέπει να έχουμε ρύθμιση τελείως ε, ε, στεγανή. Υπάρχουν κάποιες ε, ε κινητές μονάδες μέτρησης, σταθμοί, που τα λεγόμενα πάμ. Ε, που έχουν όμως ε, δυνατότητα σφάλματος 20 με 40%. Ε, υπάρχει αυτό. Ναι, υπάρχει θέμα με την ακρίβεια ή την ανακρίβεια των μετρήσεων. Τώρα λίγο πάνω, λίγο κάτω, πάντως προβλήματα υπάρχουν. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να είναι μία δοκιμή στην οδήγηση και να παίρνουμε αυτά τα στοιχεία, αλλά να κάνουμε δέκα δοκιμέ με οδήγηση, πραγματικέ συνθήκες, και να παίρνουμε το μέσο όρο να το ανάγουμε για να έχουμε έτσι, γερά στοιχεία. Τεχνικά μέχρι πότε θα χρειαστεί, πιστεύετε, η ε, ανακρίβεια στις μέτρες να είναι 30%, να μειωθούν στο 5%. Δηλαδή μέχρι πότε θα περιμένουμε για να γίνει αυτό. Το 2017 είπατε θα γίνουν τα ήδη τα ηλεκτρονικά αυτά συστήματα. Είναι ε, ρεαλιστικό. Είναι ρεαλιστικό. Γίνονται συνεχώς βελτιώσεις στις ε, διαδικασίες και τις μεθόδους μέτρησης είναι κοντά χρονικά. Εγώ δεν είμαι τώρα τεχνικός για να σας απαντήσω τα τεχνολογικά και να τα πάρετε και τις μετρητής αυτά που θα σας πω. Ναι, μια ερώτηση συμπληρωματική αφού μας επενέσατε τώρα τόσο πολύ την νομοθεσία του 2007. Η οργάνωσή σας τότε συμμετείχε στη διαβούλευση η Deutsche Umwelthilfe. Κάνατε γνωμοδοτήσεις, ελήφθη αυτή η υπόψη Τώρα πρέπει να γυρίσω σπίτι μου και να το ψάξω, γιατί τότε ακόμα δεν ήμουν ε, σε συγκεκριμένο τμήμα. Ωραία, γραπτό να μας απαντήσετε, λέει ο κύριο Γκέρκ. Ωραία. Η κυρία Σάλτεμο. Ευχαριστώ πολύ. Επανειλημμένα και στη γραπτή σας απάντηση, αλλά και σήμερα, είπατε ότι έχετε θίξει τα προβλήματα που υπήρξανε όσον αφορά τη διάφορα των αποτελεσμάτων ε, από το εργαστήριο και υποπραγματικές συνθήκες ε, και είχατε και υποψίες ε, σχετικά με το χάσμα αυτό, αλλά δεν λάβατε σαφή απάντηση από τις αρχές της Γερμανίας. Η ερώτηση μου λοιπόν είναι, Υπάρχει ανάγκη μια κυβερνητική οργάνωση όπως είναι η δική σας να έχει άλλα εργαλεία θα μπορούσαμε να ενσωματώσουμε στο σύστημα ώστε ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει ω παρατηρητέ ε, να λαμβάνουν πιο σαφεί απαντήσει από τι αρχέ. Στο παρελθόν έχουμε θέσει ερωτήματα στις αρχές. Θα τα πω γερμανικά. Στο, παρελθόν Είχαμε βασίσει τα αιτήματά μας ε, στον νόμο για την ενημέρωση σχετικά με το περιβάλλον που υπάρχει στην νομοθεσία μας. Υπάρχει όμως εδώ η δυνατότητα από τις επιχειρήσεις ε, να πούν ότι αυτό είναι ε, εμπιστευτικό και γι' αυτό πολύ συχνά λαμβάνουμε έγγραφα όπου τα μισά να είναι ε, σβησμένα, να μην φαίνεται το κείμενο. Θα θέλαμε λοιπόν να μπορούμε να ζητούμε άμεση δημοσίευση των στοιχείων και πλήρη δημοσίευση και να λαμβάνουμε τα δεδομένα που, είναι, ε, που σχετίζονται με την επανάληψη, που θα είναι χρήσιμα κατά την επανάληψη μια δοκιμή. Νομίζω ότι έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά πώς θα μπορούσαμε στο σύστημα να ενσωματώσουμε, πώ να το πω, περισσότερη καχυποψία. Όταν υπάρχουν δηλαδή ε, στοιχεία που φαίνονται περίεργο, όταν υπάρχει διαφορά στι δοκιμέ από το εργαστήριο και στι δοκιμέ υπό πραγματικές συνθήκες πώς ε, μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό ώστε να ε, ε, υποψιαστούν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ή οι αρχές μας ότι κάτι πάει στραβά. Έχετε κάποια πρόταση για το πώς μπορεί αυτό να γίνει με καλύτερο τρόπο. πληροφορίες που λαμβάνει κανείς από άλλες πηγές να μπορούν να υποβληθούν ε, στις αρχές και να υπάρχει μηχανισμός ώστε να ελεγχθούν τα στοιχεία αυτά. Και αυτό ισχύει και σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, όταν ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνονται πληροφορίες ε, ότι υπάρχει ασυμφωνία στοιχείων, να ενεργήσουν και να υπάρξει έκθεση παρακολούθησης, ώστε να υπάρχει διαφανής τεκμηρίωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία κλουνέ. Um, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ κύριε Σάρ. Και εγώ. Σχετικά με τα, τις δοκιμές RDE και τις υπόλοιπες μορφές ελέγχου και δοκιμών. Θα πρέπει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία, ακόμα είναι πρόωρη κάποια κρίση. Ελπίζουμε το σύστημα να είναι αρκετά σταθερό στο μέλλον και σοβαρό. Λέτε ότι υπάρχουν πιθανότητες και στα πλαίσια του RDE να υπάρξουν ορισμένες μετατροπές και ότι δεν φαίνεται να υπάρχει ένα ικανοποιητικό επίπεδο, αλλά υπάρχει η απέτηση για νέες τεχνολογίες στο μέλλον. Ξέρω ότι απαντήσατε σε αυτό το σχόλιο προηγουμένως. Έχετε λοιπόν κάποια ερωτηματικά σε σχέση με το πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία του RDE και πώς θα εκφραστείτε γύρω από αυτό, τι ακριβώς θα θέλατε να δείτε να γίνεται, πώς θα εκφράσετε τις ανησυχίες σας γύρω από το RDE. Κοιτάξτε, δεν έχει κλείσει το πρότυπο ακόμα. Υπάρχουν αρκετές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν. Το πώς, σαν παράδειγμα, θα προσμετρώνται τα σωματίδια. Τι είδους αυτοκίνητα θα επιλέγονται. Ε, πώς μπορούμε να αποφύγουμε προετοιμασμένα σε εισαγωγικά αυτοκίνητα. Πρέπει να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να βελτιώνει το σύστημα σε συνεχή βάση. Νομίζω ότι οι περισσότερες γνώσεις γύρω από τα τεστ αυτά ε, θα προέλθουν μέσω της χρήσης, όπως είπε ο κύριος Γκίζικε η αβεβαιότητα σχετικά με τις μετρήσεις. Πώς θα μειωθεί στο μέλλον η αβεβαιότητα αυτή. Πώς μπορούμε να διευρύνουμε ακόμα περισσότερο το πλαίσιο έτσι ώστε να αποφεύγουμε κάποιες ειδικέ προετοιμασίες στα συγκεκριμένα υποδοκιμήν αυτοκίνητα για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων των αυτοκινήτων. Πιστεύετε επίσης ότι πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και όσο προχωράει η τεχνολογία να μπορούμε να προχωρούμε και εμείς σε τέτοιες αλλαγές, λέει η κυρία Κλούν. Μια άλλη ερώτηση τώρα, πάντα από την κυρία Κλούν. Ένα ρυθμιστικό ευρωπαϊκό σώμα αντίστοιχο με το αμερικανικό θα βελτιώσει την κατάσταση σε σχέση με την αξιοπιστία των δοκιμών. Βλέπουμε τις διαφορές ιστορικά ανάμεσα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Η σύγκριση αυτή μπορεί να βοηθήσει εσάς και τα αιτήματά σας. Οι Αμερικανικές αρχές στάθηκαν στο παρελθόν πιο περίεργες θα έλεγα και γι' αυτό κατέληξαν και σε πρακτικές καλύτερες από τις αντίστοιχες της ευρωπαϊκές. Έθεσαν τις σωστές ερωτήσεις στο σωστότερο χρόνο. Επόμενη ομιλήτρια. Η κυρία Ρεβό. Είπατε ότι είναι δυνατόν ε, να γίνουν σεβαστοί οι κανόνες χωρίς να ληφθεί υπόψη ο παράγων της συμβατότητας. Είναι μια μακρά συζήτηση λέει η βιομηχανία όμως και πιστεύει ότι για να περάσει κανείς στο πεδίο ακριβώς της συμβατότητας που θα πρέπει να γίνεται σεβαστό απαιτείται χρόνος. Εσείς υποστηρίζετε ότι τεχνολογικά δεν τίθεται θέμα. Πώς θα το κάνετε αυτό. Θα ήθελα να μάθω επίσης με ποιο τρόπο και πότε εσείς ανοιχνεύσατε για πρώτη φορά τα μηχανήματα αυτά ή καλύτερα τους μηχανισμούς παραπλάνησης και θα επανέλθω. Ευχαριστώ πολύ. Την απάτη Πρόσφατα την ε, αποκαλύψαμε και στο Opel Zafira που είχαμε την υποστήριξη και των ειδικών ε, του λογισμικού ε, και ένας ειδικό που κατάφερε να διαβάσει τα αποτελέσματα και να τα συνδέσει με το λογισμικό και να τα συγκρίνει. Αποτελέσματα στο εργαστήριο και στο δρόμο. Είχαμε τις αποδείξεις. Στο παρελθόν λέγαμε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει τέτοια συσκευή που διακόπτει τη λειτουργία ένας τέτοιος συντελεστής ε, ε, συμμόρφωσης όπως αποφασίζεται δεν είναι απαραίτητος γιατί υπάρχουν δοκιμές υποχρεωτικές για τα οχήματα και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και αποδεικνύουν την πλήρη συμμόρφωση ήδη. Δεν χρειάζεται να αλλάξει. Η οδηγία για τον τύπο Euro 5 ε, και Euro 6 του κινητήρα είναι το 2007. Στο παρελθόν υπήρχαν κάποιες εκτιμήσεις ε, που τόνιζαν την τεχνική και την οικονομική δυνατότητα. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα νομοθεσίας. Αυτά ε, υπάρχουν. Ευχαριστώ. Στο τέλος της απάντησής σας υπαριθμών 13 λέγεται ότι λόγω των νόξ υπήρξαν ε, χιλιάδες ε, επιπλέον θάνατοι. Μπορείτε εσείς να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις των νόξου στο ανθρώπινο σώμα, στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό που εννοούσα είναι από το διοξίδιο του αζότου, το οποίο είναι ρυθιστικό και ε, ε, επιβαρύνει τους βλενογόνους, ε, τα αισθητήρια όργανα, τους πνεύμονες κτλ. Αυτό το δείχνουν πολλές μελέτες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος στα τέλη του περασμένου έτους έχει υπολογίσει ότι για τη Γερμανία τουλάχιστον οι πρόοροι θάνατοι είναι πάνω από 10.000 και στην Ευρώπη 72.000 για τους οποίους κατηγορείται αυτό. Ευχαριστώ κύριο Στούρμες. Ευχαριστώ πολύ. Εμένα δεν με εκπλήσει που το ήξεραν το Φεβρουάριο 2011 υπάλληλοι των Υπουργείων στη Γερμανία, γιατί από τον Νοέμβριο του 2010 υπήρξε μια κρίσιμη ε, συνάντηση 200 μέτρα από εδώ, στο Μπορσέτ, το κέντρο συνεδριάσεων, όπου το κοινό κέντρο ερευνών επιτέλους δημοσίευσε στους εθνικούς ε, εμπειρογνώμονες και παρουσίασε τα πορίσματα, ενώ είχε εμποδιστεί στο παρελθόν το Νοέμβριο 2010 ήταν ε, η χρονική έτσι, στιγμή που μετά από χρόνια ολιγορίας και ε, είχε την ευκαιρία το Κοινό Κέντρο Ερευνών να τα παρουσιάσει στους εθνικούς εμπειρογνώμονες. Άρα φυσικά και το ήξεραν τα Υπουργεία. Αυτό που βρίσκω τώρα ενδιαφέρον μεταξύ Γερμανίας και Ευρώπης. Καλά, εσείς πιστεύετε πραγματικά ότι δεν υπάρχουν πρακτικά στο Υπουργείο από τη δική σας ε, συνεδρίαση, αυτό θυμίζει και μυρίζει αυτά που συμβαίνουν εδώ. Εγώ που τη ξέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, στο εσωτερικό της έχει συστήσει ομάδα εργασίας που αντιμάχεται τη δική μας επιτροπή και φιλτράρει, διηθεί εκεί σε πολύ υψηλό επίπεδο τα mail που θα πάρουμε εμείς ή που δεν θα πάρουμε. Δεν είναι το παρόντος. Ε, πραγματικά εσείς λέτε ότι δεν κρατήσανε πρακτικά στη συνεδρίαση αυτή στο Βερολίνο που είχατε, μα τα διαβάσαμε στον τύπο. Αυτοί πάντα κρατάνε πρακτικά σε τέτοιου είδου συνεδριάσει. Πώ χαθήκαν αυτά. Τώρα εγώ μόνο εικασίε μπορώ να σα πω. Δεν ξέρω ε, τι θεωρώ χειρότερο το να μην υπάρχουν πρακτικά ή να υπάρχουν πρακτικά τα οποία έχει δει στο κοινοβούλιο και δεν του δίνονται. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να εκτιμήσω τι ισχύει τουλάχιστον η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία επόνταρε πάρα πολύ στον διζέλ τα τελευταία χρόνια με γενναία υποστήριξη της πολιτικής, είτε με φορολογικές ελαφρύνσεις, είτε άλλα κίνητρα. Και οι οριακές τιμές επίσης δεν είναι ίδιες με αυτές που έχουμε για τα βενζινοκίνητα. Και εδώ ε, είναι προνομιούχα τα ντίζελ. Και η τήρηση των ορίων δεν είναι κάτι το ανώδυνο. Είναι μια τεχνολογία πάρα πολύ περίπλοκη και εγώ δεν είμαι μηχανικός, δηλαδή δεν ξέρω αυτά τα πράγματα, που συνδέεται όμω και κάποιο κόστο η τήρηση αυτών των ορίων. Και γίνονται και επενδύσει εκεί προφανώ. Ο κύριο Τούρμες, η εκπρόσωπο του Κοινού Κέντρου Ερευνών, η κυρία Ελκουντάιρη, η οποία ήρθε και μα μίλησε, ισχυρίζεται στην απάντησή της ότι ουδής έθεσε το θέμα στο κοινό και έδρο και ερευνών για τις συσκευές Το Ρώτησε ο Σεπ Ντάνς και, και εκείνη απάντησε ρητά και κατηγορηματικά όχι. Εσείς το πιστεύετε αυτό, ότι από το 2007 που έγιναν οι δοκιμές, το 1900 98 ξέραμε ότι υπήρχαν στα φορτηγά τέτοιε συσκευέ ε, εξαπάτηση. Δεν του είχε περάσει καν από το μυαλό ότι μπορούν να πάνε και στα γεωταχεία αυτά τα πράγματα, οι παράνομε πρακτικέ. Όχι. Εντάξει, σαφή απάντηση. Ευχαριστώ κύριε Τούρμε. Αν υπάρχει στο ιστορικό τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιεπιτροπή στη δικιά μα, να μα το πείτε. Υπάρχει αντιέμιση δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι τιμή μας δεν πρόκειται να μας αποτρέψει αυτό να προχωρήσουμε στο βάθος της συζήτησης και της εξέτασης. Ο κύριος Χένκελ. Στην απάντησή σας υπαριθμών 10, στην ερώτηση 10 δηλαδή, λέτε ότι γίνονται τυχαίοι έλεγχοι δειγματοληπτικοί και με διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά. Από την άλλη, είναι επίσης σαφές ότι υπάρχουν και ακραίες ε, συνθήκες που δεν επιτρέπουν καθόλου να τηρούνται ε, αυτά τα όρια. Ποιες είναι αυτές οι ακραίες συνθήκες. Ακραίες συνθήκες, ας πούμε, μπορεί να είναι ακραία επιτάχυνση ή ακραίες θερμοκρασίες, κυρίως προς τα κάτω, πολύ ε, χαμηλές θερμοκρασίες οι συνθήκες δεν είναι γνωστές εκ των προτέρων, αλλά κυμαίνονται. Δεν εννοώ ότι κάνουμε δοκιμές όπου συναθρίζουμε όλες τις ακραίες μεταβλητές και κάνουμε εκεί τη δοκιμή. Τις αλλάζουμε, λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία αυτά στο πλαίσιο ε, της κανονικής συμπεριφοράς οδήγησης. Σε όλες αυτές τις δοκιμές λοιπόν που κάνατε, σα πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι μπορεί να υπάρχει και διαφορετική ποιότητα δίζελ, το πετρέλαιο να φταίει δηλαδή για τα καυσαέρια. Μπορεί στα πλαίσια των απαιτήσεων να υπάρχει διαφορά από πετρέλαιο σε πετρέλαιο που να επηρεάζει και τις εκπομπές καυσαερίων, αλλά δεν εξηγούν αυτές οι μεγάλες διαφορές που βρήκαμε στις μετρήσεις μας. Και τελευταία ερώτηση. Με βάση τα όσα σήμερα δηλώσατε εδώ, δημιουργείται η εντύπωση ότι θέλετε να καταργήσετε την πετρελοκίνηση στα αυτοκίνητα, τον ντίζελ ε, Ισχύει αυτό, όχι δεν ισχύει. Αν θέλουμε να είναι καθαρό το ντίζελ και το αυτοκίνητο ντίζελ, για να κυκλοφορεί μια χαρά αν καθαρίσει. Εμείς δεν είμαστε ούτε υπέρ ούτε κατά του δίζελ, ούτε υπέρ κατά της βενζίνης ή άλλου καυσίμου. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι με τρόπο τεχνολογικά ουδέτερο να έχουμε το αποτέλεσμα που να είναι καθαρά αυτοκίνητα που να κυκλοφορούν στους δρόμους. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάντενμπαχ. Ευχαριστώ πολύ που βρήκατε χρόνο για να συζητήσετε μαζί μας εντατικά. Θέλω να συνεχίσω από μια ερώτηση που έκανε προηγουμένως η Κριστίν Ρεβονταλόν και να σας πω ότι έγραψε μια αυστριακή ε, εφημερίδα. Ένας έμπορος αυτοκινήτων, Καρλ Όπμαν, ε, λέει ότι θα προσφύγει γιατί μας κάνετε ζημιά. Και λέει ε, ότι αυτό δεν, δεν ζημίωσε κανένα και ο κόσμος δεν αγόραζε τα ντίζελ επειδή εκπέμπουν λιγότερα καυσαέρια. Δηλαδή, αυτό εσείς πώς το βλέπετε. Το βλέπετε να το λένε και οι γερμανικές κρατικές αρχές. Ότι πρόκειται για μια διοικητική παράβαση. Ωραία δεν τηρήσαμε την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είχαν επίγνωση, έχουν επίγνωση αρμόδιο ότι αυτή η νομοθεσία ε, είχε και κάποιο στόχο να μειωθούν οι εκπομπές καυσαερίων έτσι ώστε πρώτον να προστατεύεται η δημόσια υγεία και δεύτερον το περιβάλλον ή να είναι η ειναι όσο γίνεται μικρότερη. Μιλήσατε για 10.000 πρόωρους θανάτους στην ε, Γερμανία, 72.000 στην Ευρώπη, πρόωροι θάνατοι έτσι από αυτά τα καυσαέρια, από εκπομπές ε, ε, οχημάτων. Ε, με κάποια εγγυακά νοσήματα, αναπνευστικά και πάει λέγοντας. Είναι τεράστια η ζημία και στα δημόσια οικονομικά πέρα από τη δημόσια υγεία. Αυτή τη διάσταση την ξέρουν, έχουν επίγνωση οι αρχές και για λόγους χρονικούς να συνεχίσω με τη δεύτερη ερώτηση. Έχω την αίσθηση ότι κατά τη διάρκεια των δικών σας δοκιμών και της ε, δημοσιοποίησης ε, του προβλήματος Ετεχθήκατε κρούσεις από κάποιους κατασκευαστές αυτοκινήτων και σας εμπόδισαν να τα κοινοποιήσετε αυτά στο ευρύ κοινό. Ισχύει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το παράδειγμα που μόλις αναφέρατε αποτελεί πολύ ακραία διατύπωση. Δεν συναντήσαμε κάτι τέτοιο στις ε, γερμανικές αρχές. Υπάρχουν αυτές οι δύο προκλήσεις, από τη μία η διασφάλιση της κινητικότητας, και ε, το ότι λαμβάνουμε υπόψη ότι σημαντικό ε, προϊόν για τους ε, Γερμανούς κατασκευαστές αυτοκινήτων είναι τα αυτοκίνητα που κινούνται με ντίζελ. Από την άλλη θέλουμε να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων. και μάλλον ε, δεν ε, είχαν τόση αποφασιστικότητα οι γερμανικές ε, αρχές να προστατεύσουν την υγεία όσον αφορά τις, τα γερμανικά αυτοκίνητα. Η εταιρεία Daimler πριν ε, τη δημοσίευση στοιχείων τους ε, μας είπαν ότι θα θεωρήσουν ότι είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε οικονομική ζημία που θα υποστούν ε, από τη δημοσίευση των στοιχείων αυτών. Μας απαγόρευσαν επίσης να δημοσιεύσουμε την σχετική επιστολή του δικηγόρου τους. Το κάναμε αυτό και υπήρξε κατόπιν δικαστική απόφαση. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριο Σφέτερλε. Α, όχι, συγγνώμη. Ο κύριος Κερμπράντη. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, αν ε, ένας καθηγητής δώσει στον μαθητή, τον σπουδαστή, τις ερωτήσεις του διαγωνισμού εκ των προτέρων, ξέρουμε ότι ο μαθητής θα μάθει μόνο τα συγκεκριμένα θέματα. Το ίδιο γίνεται και στις δοκιμές αυτοκινήτων, διότι η βιομηχανία γνωρίζει τι μορφή έχουν οι δοκιμές. Μάλιστα συμμετέχουν ε, στην εκπόνηση των δοκιμών. Πώς βλέπετε εσείς τη διαδικασία αυτή και βρίσκεται σωστή τη σύγκριση που κάνω με τον ε, καθηγητή και τον μαθητή και γίνεται κάτι παρόμοιο με άλλα καταναλωτικά αγαθά. Συμμετέχουν οι ε, κατασκευαστές εξίσου στις ε, δοκιμές ή για παράδειγμα στα ψυγεία. Να απαντήσω πρώτα στη δεύτερη ερώτησή σας. Νομίζω πως ναι, αλλά δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένο παράδειγμα. Για παράδειγμα στον τομέα της ψήξης ε, ή του κλιματισμού. Πολλές ε, λεπτομέρειες ε, θεσπίζονται όχι από τον νομοθέτη, αλλά από πρότυπα DIN, DIN τα οποία τα καθορίζει η ίδια η βιομηχανία. Όσον αφορά το παράδειγμα σας ε, του δάσκαλου και του μαθητή, είναι απόλυτα σαφές και συμφωνώ. Από την άλλη, Εάν συμφωνήσουμε ότι μια συγκεκριμένη δοκιμή αποτελεί και τη βάση για την πιστοποίηση, θα πρέπει να είναι σαφής η δοκιμή, ώστε να είναι πιο εύκολο όχι μόνο για τον ε, κατασκευαστή, αλλά και για ε, τον φορέα δοκιμών. δύσκολο είναι να συμπεριλάβει κανείς σε μια ευρύτερη ε, οπτική που έχει να κάνει με την πραγματική χρήση του προϊόντος. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι ε, υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Νομίζω ότι έτσι θα πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Η ε, Γκρέφιν Φοντούν και Ευχαριστώ πολύ. Πήρε ένα ταξί σήμερα στις Βρυξέλλες και ήταν ηλεκτρικό το αυτοκίνητο και ο οδηγός μου είπε ότι πέρασε από το πετρελαιοκίνητο στο ηλεκτρικό εδώ και 9 μήνες. Πριν 9 μήνες είχαν 9 ηλεκτρικά αυτοκίνητα και σήμερα 80. Um, Ποιο είναι το μέλλον λοιπόν της πετρελαιοκίνησης και ποιες είναι οι τεχνικές δυνατότητες. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι σε θέση να στραφεί στο μέλλον σε σχέση και με τις εκπομπές και με την αποδοτικότητα στον τομέα της κατανάλωσης. Ποια είναι τα βασικά εμπόδια στο, για το μέλλον για την πετρελαιοκίνηση υπάρχει δυνατότητα μείωσης των περαιτέρων. Υπάρχει τεχνολογία στην αγορά και νομίζω ότι κάθε χρόνο τα αυτοκίνητα της πετρελαιοκίνησης είναι καθαρότερα και δεν υπάρχει λόγος να μην χρησιμοποιείται στο μέλλον. Υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει και καλύτερη επίδοση στον τομέα ε, της, ε, των εκπομπών, αλλά αυτό σημαίνει προσπάθεια παρέμβασης και σε σχέση με τη λειτουργία της μηχανής και με το βάρος του οχήματος. Θα δούμε αν βασικός στόχος είναι η πλήρης ηλεκτροκίνηση. Αυτό έχει κάποιο νόημα. Αν θέλουμε εμείς να πετύχουμε τους στόχους μας θα πρέπει μέχρι το 2030 να έχουμε μηδενικές εκπομπές σε ορισμένα ίχνοστοιχεία. Για τις υπάρχουσες τεχνολογίες λέει η κυρία Τούν. Ποιο είναι το βιομηχανικό κόστος ε, για τις εταιρείες. Υπάρχουν τεχνολογίες όπως είπατε για τη μείωση και των NOx, αλλά αυτό το επιπλέον κόστος. Θα βοηθήσει, θα επιτρέψει την παραγωγή των νέων αυτών πετρελαιομηχανών ή μήπως η χρήση αυτών των μικρού μεγέθους ε, ε, κινητήρων ε, είναι κάτι το πάρα πολύ ακριβό και τίθενται θέματα ανταγωνιστικότητας. Σύμφωνα με την άποψή σας λοιπόν υπάρχουν συστήματα και δυνατότητες που να επιτρέπουν την πρόοδο. Κοιτάξτε, για τα μικρά αυτοκίνητα ίσως να είναι πολύ ακριβή η τεχνολογία υπάρχει από την ICCT μια, ένας πίνακας σύγκρισης κόστους ανά είδος καυσίμου. Θα έχουμε και γραπτέ ερωτήσει, οπότε μπορείτε εκεί να υποβάλλετε πλέον ερωτήσει. Ο κύριο Σούλσε, ε, κύριε Ζάρ, σα ευχαριστώ πολύ που βρίσκεστε εδώ σήμερα το πλεονέκτημα όταν παίρνει κανείς το λόγο τελευταίο είναι ότι έχουν ήδη απαντηθεί ε, πολλές από τις ερωτήσεις ε, που ήθελα να θέσω. Αλλά είπατε ότι μπορείτε να κάνετε εσείς μόνο δειγματοληπτικούς ελέγχους. Πώς επιλέγετε λοιπόν ε, τα αυτοκίνητα που ελέγχετε ή υπάρχει κάποιος μηχανισμός για την επιλογή ή κάποια μέθοδος. Με φορητές συσκευές ελέγχουμε ε, τα 30 πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στις ε, νέες άδειες κυκλοφορίες που έχουν εκδοθεί. Σκεφτήκατε ποτέ να εξετάσετε αυτοκίνητο το Ιώτα παρότι δεν ε, βρίσκεται στα 30 πρώτα. Ναι, το σκεφτήκαμε. Πέρα από αυτά τα 30 πιο δημοφιλή αυτοκίνητα, όπου πολύ πιθανό να υπάρχει και ένα Toyota, θα εξετάσουμε μοντέλα ώστε να καλύψουμε όσο γίνεται πιο μεγάλο ε, εύρος αυτοκινήτων που χρησιμοποιούνται από Γερμανούς οδηγούς. Ο κύριος Σούλσε. Ε, η εντύπωσή μου είναι ότι δεν σας πήραν απόλυτα στα σοβαρά οι αρχές. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι, για παράδειγμα, έχετε λάβει χρηματοδότηση από την Toyota. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Είναι πολύ διαφανή τα έσοδά μας. Εδώ και πολλά χρόνια είναι γνωστό ότι λαμβάνουμε οικονομική υποστήριξη από, μέλη, από, από, από τη βιομηχανία. Από εκεί και πέρα δεν είμαστε οι μόνοι που επισημάναμε το πρόβλημα απέναντι στις αρχές. Έχω ακόμα δύο ερωτήσεις. Είπατε ότι είναι απόλυτα διαφανής η οργάνωσή σας. είσαστε διατεθειμένοι να δημοσιεύσετε τη συμφωνία με την Toyota. Είπατε ότι ε, λαμβάνετε χρήματα, αλλά αυτό δεν λέει πολλά. Και μία τεχνική ερώτηση. Κάνατε πριν τη σύγκριση των ζώνων ασφαλείας με τις διατάξεις αναστολής. Δηλαδή, ας φανταστούμε ότι οι ζώνες ασφαλείας δεν λειτουργούν ε, από κάποια ε, θερμοκρασία και πάνω. Ε, εγώ ως άνθρωπος της τεχνολογίας εκπλήσωμαι από μια τέτοια δήλωση. Δεν ε, συνέκρινα τις ζώνες ασφαλείας. Απλά ε, ανέφερα ότι το in normal use υπό συνθήκες, ε, η φράση αυτή υπάρχει στα πρότυπα και για τα μεν και για τα δε. Θα απαντήσετε και στην προηγούμενη μου ερώτησή σας. Πολλές ερωτήσεις, Πολλές ερωτήσεις κάνετε. Έχετε μια συμφωνία με την Toyota, θα την κοινοποιήσετε. Όχι. Μπορώ να σας ενημερώσω, αν θέλετε, Όχι, μου αρκεί η απάντηση, Κοιτάξτε, δεν εξετάζουμε, δεν ανακρίνουμε τη ΜΚΟ σήμερα. Τελευταίος ο κύριος Ντάνς. uh... Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Μέχρι στιγμής ήταν πάρα πολύ χρήσιμες. Είστε κατηγορηματικοί λέγοντας ότι η νομοθεσία είναι εντάξει, είναι σαφής. Ε, το πρόβλημα είναι η ερμηνεία που υπολείπεται, για να το πω έτσι ήπια. Δεν πω τίποτα πιο χοντρό. Και ότι υπήρξε και παράνομη συμπεριφορά στι συσκευέ εξαπάτηση. Τι γίνεται τώρα με τη νέα νομοθεσία για τις νέες δοκιμέ και τη νέα τεχνολογία που υπάρχει. Είπατε ε, ότι η δυσκολία με το, το PEMS στις χωρητές συσκευές είναι ότι ε, αλλάζει το κέντρο βάρους ε, προς τα πίσω στο αυτοκίνητο. Και τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή. Τι θα συστήνατε στο Κοινοβούλιο για να μην υπάρχουν παραθυράκια στη νέα νομοθεσία. Κοιτάξτε. να αποφευθεί η δοκιμή πούμε, του χρυσού αυτοκινήτου ένα, που να είναι ένα πρωτότυπο αλλά είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο να κυκλοφορεί στους δρόμους και να συγκριθούν τα αποτελέσματα με δοκιμές άλλων αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Δεν υπάρχει σύστημα κυρώσεων, τουλάχιστον στη γερμανική νομοθεσία. Αυτό θα μπορούσε να μας βοηθήσει να οριστεί ένα πλαίσιο για το τι επιτρέπεται και τι όχι. Και να υπάρχουν συγκρίσιμοι μηχανισμοί, όπως στις ΗΠΑ. Αυτά τα δύο. Και φυσικά διαφάνεια και δημοσίευση των στοιχείων. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ ολοκληρώνεται η πρώτη ακρόαση σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Σάρ για την ειλικρίνεια στις απαντήσεις σας. Θα ακολουθήσουν και οι συμπληρωματικές γραπτές ερωτήσεις προς την οργανωσή σας Deutsche Umwelthilfe. Σας ευχαριστώ και πάλι και να τα ξαναπούμε. Στο καλό να πάτε. Can I, can I please ask that, Χούντεμαν και Σαμπίντο, Okay, I would like to welcome the guests of our second hearing of today, Mr. Pasqualido. Να, να υποδεχθώ τους κυρίους Χόιντεμαν και Σαμπίντο. Σας ευχαριστούμε για την ε, παρουσία σας εδώ. Θα δώσετε απαντήσεις. Έχετε 10 λεπτά και οι δύο Corporate Europe Observatory, CEO, είναι μια ομάδα η οποία θέλει να υπογραμμίσει και να αποκαλύψει την πλεονεκτική θέση και πρόσβαση σε ενημέρωση και πληροφορίες που έχουν οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, λέει ο κύριος Σαμπίντο, ελπίζω να βοηθήσουμε από πλευράς μας. Όπως είπαμε, εμείς είμαστε μια διερευνητική ε, οργάνωση που οργανώνει εκστρατείες ε, για την ε, πρόσβαση των μεγάλων επιχειρήσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Εμείς δεν είμαστε τεχνική οργάνωση, ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων στην περίπτωση κατά την οποία δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε τεχνικές ερωτήσεις. Νομίζω ότι όπως η κυρία Σάρ θα μπορούσε να δώσει καλύτερες απαντήσεις. Η ανάλυση μας δείχνει ότι υπάρχει έντονο λόμπινγκ από την αυτοκίνητο βιομηχανία και από τις Βρυξέλλες και σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν στενές επαφές με αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Υπάρχουν μαθήματα τα οποία μπορούμε να μάθουμε να βελτιωθεί η διακανονιστική διαδικασία. Ήδη στο τέλος Ιανουαρίου δημοσιεύσαμε το πρώτο έγγραφο που βασίζεται σε σχέση με τις θετικές απαντήσεις σε πρόσβαση για προσβάσεις σε ενημερώσεις που είχαμε καταθέσει ήδη από το 2015. Στείλαμε τις ερωτήσεις και στην ΑΣΕΑ, την Ομοσπονδία, την Ευρωπαϊκή των Αυτοκίνητων Βιομηχανιών και την Ευρωπαϊκή Ένωση η ε, επιστολική αλληλογραφία η οποία δημοσιεύθηκε δείχνει ότι οι διαδικασίες ε, είχαν ε, γίνει δεκτές σε επίπεδο ευρωπαϊκό τον Οκτώβριο. Η αυτοκίνητο-βιομηχανία πλάκη στη διαδικασία συγγραφής της νομοθεσίας. Εκεί που επέμενε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν υπέκυπτε το λόμπι υπήρξε ιδιαίτερα ιστηρό προσπάθησαν να αποδυναμώσουν την πρόταση, να καθυστερήσουν ε, και επίσης ε, δημιούργησαν προβλήματα σε σχέση με τους, ε, με τους παράγοντες συμβατότητας ή παράγοντες συμμόρφωσης. Χρησιμοποίησαν τα τεχνικά προβλήματα για να υπονομεύσουν τις προτινόμενες διαδικασίες του κύκλου δοκιμών ε, προσπάθησαν να επηρεάσουν το τι σημαίνει κανονικός ρυθμός οδήγησης έτσι ώστε ε, να υπάρξουν πιο ευνοϊκές απαντήσεις για αυτούς όπως σαν παράδειγμα οι κινήσεις του κινητήρα με χαμηλές θερμοκρασίες και γενικά να οδηγήσουν σε κανόνες οι οποίοι να θεωρούνται εύκολοι για την βιομηχανία και να μπορέσει να είναι συμβατά τα αποτελέσματα σε σχέση με τις απαιτήσει παρά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην υγεία. Υπήρξε πολιτικοποίηση λοιπόν της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης και δείχνει επίσης και την έλλειψη της αντίστοιχης εμπειρογνωμοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξαν και ολόκληρα κράτη-μέλη που προσπάθησαν να επιβραδύνουν τις διαδικασίες, χρησιμοποίησαν και τεχνικά προβλήματα, η ΑΣΕΑ σαν παράδειγμα η Ομοσπονδία των Αυτοκίνητων Βιομηχανιών ε, μία εβδομάδα πριν κάνει τις προτάσεις της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε τις δικές της προτάσεις τεχνικές προσπαθώντας να προκαλέσει κολυσιεργία. Ε, για την αποδυνάμωση των παραγόντων συμβατότητας ή ε, συμμόρφωσης χρησιμοποιήθηκαν και απειλές ότι θα κλείσουν τα εργοστάσια, θα χάσουμε θέσεις εργασίας, ύβρις, ε, απόρριψη των ε, παραγόντων που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απειλές χρήσης ένδικων μέσων ε, έτσι ώστε να αποδείξουν ότι μπορούν να υπονομεύσουν τους κανόνες αυτούς τους παράγοντες συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς τον Μάρτιο του 2015 δημοσιεύσαμε μια δεύτερη έκθεση βασισμένη σε ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε ε, που λέγει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε μια κάποια συμβιβαστική στρατηγική στον τομέα αυτό και βασιζόταν σε πληροφορίες οι οποίες προήλθαν σε επίπεδο ανεπίσημων επαφών δεν υπήρξε αναφορά σε αυτές τις επαφές σας ε, και δεν ήταν στον κατάλογο των επίσημων επαφών και ε, τα στοιχεία αυτά ήταν αντίθετα με όσα χρησιμοποιούσε μέχρι τότε η Επιτροπή. Και αυτές οι επιπλέον πληροφορίες βοήθησαν την βιομηχανία να κρατήσει μια πιο σκληρή αν θέλετε ε, γραμμή. Και δεύτερον ένας άλλος κομβικός παράγων από το, από το κείμενο το οποίο διέρευσε είναι η περιπλοκότητα της στρατηγικής που καλύπτει επαφές σε επίπεδο λήψεως αποφάσεων και εδώ στις Βρυξέλλες και σε εθνικό επίπεδο, σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο αναχώρα και στα πλαίσια μιας ολοκληρωμένης αν θέλετε και περίπλοκης στρατηγικής έτσι ώστε όταν δεν ανταποκρινόταν μόνη της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρεμβαίνουν οι χώρες. Το λόμπι αυτό εν πολλής παρουσιαζόταν κυρίως σαν τεχνικό input, πληροφόρηση και ενημέρωση την οποία είχε ανάγκη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ότι υπήρχε δήθεν κίνδυνος επικαλύψεων σε σχέση με την εμπειρογνωμοσύνη αυτή όταν εφήγονται τα συμφέροντα των βιομηχανιών. Νομίζω ότι οι ίδιες λοιπόν οι βιομηχανίες οι οποίες έπρεπε η παραγωγή τους να ρυθμιστεί παρενέβησαν για να ορίσουν το πώς θα γίνει η ρύθμιση αυτή. Τώρα συνεχίζει ο έτερος των ομιλητών ο κύριος Χέντεμαν σας ευχαριστώ πολύ. Είναι σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να, να προστατευτεί περισσότερο η λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από υπερβολική επιρροή από πλευράς ε, της βιομηχανίας αυτοκινήτων. Στις γραπτές μας ε, απαντήσεις Έχουμε προτείνει διάφορους τρόπους ε, να προστατευτεί η ποιότητα της λήψης αποφάσεών σας. Ε, αυτό συμπεριλαμβάνει την διαφάνεια στις δραστηριότητες ε, lobbying, καθώς και την επιγραμμική δημοσίευση συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων και ενδιαφερομένων κύκλων. αναφέρονται επιγραμμικά κάποια στοιχεία, αλλά αποτελούν μόλις την κορυφή του παγόβουνου και οι έρευνες μας δείχνουν ότι πολύ μεγάλος αριθμός συναντήσεων με τους λομπίστες ε, πραγματοποιείται σε επίπεδο χαμηλότερο ε, από ε, τους αξιωματούχους που δημοσιεύουν τις συναντήσεις τους επιγραμμικά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν πρακτικά των ε, συναντήσεων αυτών. Ε, μία από... Ένα από τα απογοητευτικά συμπεράσματά μας ήταν ότι πολλές συναντήσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τους λομπίστες δεν... Στις συναντήσεις αυτές δεν κρατήθηκαν πρακτικά δεν είμαστε αφελείς όσον αφορά τη διαφάνεια, δεν θα εμποδίσουμε έτσι την υπερβολική επιρροή της βιομηχανίας αυτοκινήτων, αποτελεί ένα βήμα, αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να υπάρξει σαφώς, σαφές μήνυμα από την κορυφή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει να υπάρξουν πολύ συγκεκριμένα μέτρα μεταρρύθμισης όσον αφορά τις συναντήσεις με τα λόμπι. Τρία πράγματα να αναφέρω ακόμα. Πολύ σημαντικό είναι να μειωθεί η εξάρτηση από τον ε, τομέα που θέλει να ρυθμίσει η Επιτροπή, την ε, βιομηχανία αυτοκινήτων στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει δηλαδή η Κομισιόν να έχει δική, δικούς της εμπειρογνώμονες ε, ή εμπειρογνώμονες ανεξάρτητους από τη βιομηχανία αυτοκινήτων. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τις συναντήσεις με, δια, με τους διάφορους ενδιαφερομένους. Ο πρόεδρος ε, Γιούνκερ ε, στο τέλος του 2014 έδωσε οδηγίες στους επιτρόπους, τους, ε, τους του να υπάρχει ευρεία εκπροσώπηση όσον αφορά τους ενδιαφερομένους που συναντούν. Αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί και να καλύπτει όλους τους αξιωματούχους της Κομισιόν. Υπάρχουν πολύ συχνέ ε, και πολύ στενέ επαφές ε, ανάμεσα σε λομπίστε τη ε, βιομηχανία αυτοκινήτων και υπαλλήλου τη Κομισιόν. Πιστεύουμε λοιπόν ότι χρειάζεται μια πιο επίσημη προσέγγιση και πιο σαφείς κανόνες για τις επαφές αυτές. Υπάρχουν σημαντικές αρχές στις οδηγίες για τι διαβουλεύσει τη Κομισιόν και στις οδηγίες ε, που δίνει η Κομισιόν στους υπαλλήλους της, αλλά είναι υπερβολικά γενικοί οι κανόνες αυτοί και υπερβολικά περιορισμένοι. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πιο σαφείς ε, και να εφαρμόζονται πιο σωστά. Υπάρχουν ε, παρόμοια προβλήματα και σε εθνικό επίπεδο. Τέτοιες μεταρρυθμίσεις λοιπόν θα πρέπει να συζητηθούν και σε εθνικό επίπεδο. Θα κλείσω εδώ και περιμένω να απαντήσω στις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος. Πρόσωποι των πολιτικών ομάδων για πέντε λεπτά. Ε, ερώτηση και απάντηση. Ο κύριος Χερπράντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους δυο σας για την παρουσίαση. Τώρα τι συζητάμε. Την ε, λεπτή και ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα ε, στη σωστή πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να βελτιωθεί η νομιθική μας προσπάθεια από μια και από την άλλη την υπερβολική πρόσβαση και αρνητική επιρροή έτσι, ε, στην ε, χάραξη πολιτικής και λήψη αποφάσεων. Έχω να ρωτήσω το εξή. Αν συγκρίνετε την πρόσβαση που έχει επίσημα η αυτοκινητοβιομηχανία σε σύγκριση με άλλες βιομηχανίες, υπάρχει καμιά διαφορά. Ε, ε, η οργάνωσή μας έχει κάνει μια έρευνα σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας και παντού ισχύει αυτό. Θα πρέπει να δούμε γενικότερα γιατί ισχύει αυτό. Και γιατί ιδιαίτερα αυτοκινητοβιομηχανία, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει στο εσωτερικό τη εμπειρογνώμονε με τέτοιε τεχνικέ και τεχνολογικέ γνώσει ε, που να μην εργάζονται στην αυτοκινητοβιομηχανία, δηλαδή δεν υπάρχουν ειδικοί όταν παίρνουν ε, ομάδες εμπειρογνωμόνων δηλαδή ε, και τους ε, συμβουλεύονται, άλλο ομάδα εργασίας, 66% των εκπροσώπων είναι εκπρόσωποι της βιομηχανίας και ειδικά στο σύστημα RDE, στο Real Drive Emissions είναι πολύ περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αλλά αυτό ανάγεται και σε μια πολιτική επιλογή γιατί δεν υπάρχει εσωτερική πραγματογνωμοσύνη. Ε, σε σύγκριση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα ότι αυτή τη θέση θέλουμε να έχουμε στην Ευρώπη. δεν καταλαβαίνουμε την ενδεχόμενη σύγκρουση φερόντων που μπορεί να προκύψει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος Έχουμε περιέλθει τώρα σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθούμε να ε, ε, εγγυηθούμε την ανεξάρτητη ε, πραγματογνωμοσύνη. Αυτό είναι σχεδόν αδύνατο. Ε, ακόμα και οι εγκαταστάσεις που κάνουν τον τεχνικό έλεγχο εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση των εργοστασίων δεν ξέρω, αλλού ε, σε άλλους κλάδους οι πανεπιστημιακοί οι ομάδες πολιτών ε, μπορούν να επηρεάσουν, αλλά για τις μεταφορές και ιδιαίτερα για τα αυτοκίνητα είναι πολύ λίγοι εξωτερικοί εμπειρογνώμονες που δεν εργάζονται ήδη στην αυτοκινητοβιομηχανία. Άρα τι μας λέτε τώρα ότι δεν έχουμε γνώση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τεχνογνωσία για αυτά τα θέματα και αυτό είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα, ακόμα μεγαλύτερο από την πρόσβαση της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στις γραπτές απαντήσεις σας αναφέρετε ότι από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι το Φλεβάρι του 2016 υπήρξαν 21 επίσημες συνεδριάσεις ε, της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης με την ΑΣΕΑ. Αυτό είναι σε μηνιαία βάση και παραπάνω. Τόσο συχνά συνεδριάζουν αυτοί. Είναι φυσιολογικό αυτό. Άλλοι κλάδοι της βιομηχανίας έχουν τόσο συχνές συνεδριάσεις πάνω από μία φορά το μήνα. Εγώ δουλεύω και για το κλίμα και στα, στα ορυκτά καύσιμα με τον Επίτροπο Κανιέτη συναντιούνται όντως πάνω από μια φορά το μήνα. Αλλά πέραν των επισήμων διάβλων ε, επιρροής Υπάρχουν και τηλεδιασκέψεις ε, και τα λοιπά. Στη Task Force επίσης συμμετέχουν ε, μέλη τους. Δεν είναι μόνο επίσημες συνεδριάσεις. Έχουν και άλλους διάβολους επικοινωνίας. Η Volkswagen συμμετέχει σε πέντε διαφορετικές ομάδες εμπειρογνωμόνων. Έχουν και άλλους τρόπους να βρίσκονται πέρα από αυτές τις επίσημες συνεδριάσεις. 21 συνεδριάσεις είναι αυτές που γνωρίζουμε. Μπορεί να, και δεν λέω για άτυπε, μπορεί να υπάρχουν και επίσημες που να μην δημοσιεύονται. Γιατί όταν εμείς ε, ε, ζητήσαμε στοιχεία επίσημα, ξέχασαν να μας αναφέρουν κάποιες συνεδριάσεις και στη συνέχεια τις προσέθεσαν. Υπάρχει πρόβλημα στην ε, εθελοντική διαφάνεια από πλευρά του, στην αυθόρμητη. Η αυτοκινητοβιομηχανία πραγματικά συμμετέχει πάρα πολύ στην όλη νομοθετική διαδικασία. Θα λέγατε λοιπόν ότι σε αυτές τις τεχνικές ομάδες εκπροσωπείται πιο μαζικά η αυτοκινητοβιομηχανία από άλλες ε, μορφές, άλλους κλάδους της βιομηχανίας στις αντίστοιχες ομάδες. Δυστυχώ όχι. Εγώ εργάζομαι και εγκάρσια σε ομάδε εμπειρογνωμόνων και είναι μεγάλο πρόβλημα αυτή η ανισορροπία. Και οικονομικά και πολιτικά σημαντικέ ομάδε κυριαρχούνται από ομάδες της βιομηχανία και σε επίπεδο απαρτία. δηλαδή υπερτερούν αριθμητικά. Δεν είναι ίδιον μόνο αυτό της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σάλβα, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ ε, και τους δυο σας για αυτά που μας είπατε. Όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη νέα πρόταση και ε, πλήρη για το ένα νέο πλαίσιο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και τις ανεπάρκειες που μεταξύ άλλων εσείς μας αναφέρετε. Πώς αξιολογείτε εσείς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που καταρχήν φαίνεται να είναι η πιο προηγμένη παγκοσμίω και η πιο πρωτοπόρο. Ευχαριστώ. Ποια πρόταση αναφέρεται για τις αρχές που εγκρίνουν τον τύπο για το πακέτο, αυτή η τελευταία πρόταση που έχει να κάνει τις δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες real drive emissions και όχι σε ε, εργαστήριο. Κοιτάξτε, εγώ τεχνικός εμπειρογνώμων δεν είμαι. Ε, προσωπική δουλειά έχω κάνει για να ψάξω να βρω όλα αυτά τα θέματα, να καταλάβω γιατί γίνεται όλη αυτή η πίεση και το λόμπι μήπως να ρωτήσετε τους ειδικού. Εμεί έχουμε την αίσθηση ότι οι προτάσεις αυτές είναι καλύτερες από τις προηγούμενες, αλλά κοιτάζοντας τα έγγραφα που λάβαμε και τα ε, παραθυράκια που έχουν, υπάρχουν ε, σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις. Έχω κάνει κατάλογο ολόκληρο εδώ πέρα, ε, στην αρχική μου παρουσίαση. Ας πούμε, οι θερμοκρασίες υποτίθεται ότι θα ήταν μηδέν βαθμοί και τώρα είναι τρεις. Ε, η ψυχρή εκκίνηση που είναι κάτι το τρέχουν και στις σκανδιναβικές χώρες και το χρησιμοποιούν και σε τεστ ε, στις συνθήκες ε, πραγματικής οδήγησης και τα λοιπά. Μπορεί να σας φαίνονται λεπτομέρειες, αλλά αν θρηστούν συγκεντρώνονται πολλά. Και αυτές οι τεχνικές αλλαγές χρειάζονται μάλλον έχουν μπει για να χαλαρώνουν ε, ε, οι ρυθμίσεις, να υπάρχουν παραθυράκια και να ε, μπορούν οι εταιρείε να μην τηρούν τις προδιαγραφές. Και για τον κινητήρα Euro 6 πραγματικά υπάρχουν ακόμα διαφορές ανάμεσα με το τι σημαίνει στον πραγματικό κόσμο, στην πραγματική οδήγηση και στις δοκιμές. Τώρα, αν θα υπάρχει ειλικρίνεια και διαφάνεια και παράγοντες συμμόρφωσης, έχει το 2021 η αυτοκινητοβιομηχανία θα έχει ξεπεράσει κατά 50% το όρια του κινητήρα Euro 6. Ο κόσμος θα τα γνωρίζει, άραγε μπορεί να βελτιώνονται τα συστήματα μετρήσεων και ελέγχου, αλλά ε, η αυτοκινητοβιομηχανία και τα κράτη-μέλη έχουν φροντίσει να υπάρχουν αρκετά παραθυράκια έτσι ώστε να μην στριμώχνονται. Κατά τη γνώμη σας, ποια θα ήταν η ιδανική πρόταση για να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα τα οποία, τα οποία περιγράφετε. Πιστεύετε δηλαδή ότι κάτι που θα, μια απόφαση που θα ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα ε, έχει αντίκτυπο σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορώ να ξεφύγω από τα όρια της εμπειρογνωμοσύνης μας ε, σήμερα, αλλά υπάρχουν οργανώσεις όπως η DUH και άλλες ε, που έχουν εξετάσει τέτοιες προτάσεις, αλλά οποιαδήποτε πρόταση θα πρέπει να φροντίσει ε, η βιομηχανία αυτοκινήτων ε, να συμμορφώνεται με τα όρια τα οποία θεσπίστηκαν για να προστατευτεί η δημόσια υγεία και να ε, αποτρέψουμε πρόορους θανάτους. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη συμμόρφωση και είτε το κάνουμε αυτό σε ευρωπαϊκό, παγκόσμιο ή εθνικό επίπεδο θα πρέπει να ισχύει για για όλους και θα πρέπει να φροντίσουμε να, να προστατεύεται η λήψη αποφάσεων από ε, αθεμητή επιρροή. Ευχαριστώ αν κατάλαβα σωστά. Θέλετε όχι νέο κανονισμό, αλλά καλύτερη συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό. Σωστά τα λέω. Νομίζω ότι όταν υπάρχει κανονισμός που, είναι αποτέλεσμα, που πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας δημοκρατικής διαδικασίας και είτε μιλάμε για τον ισχύοντα είτε μιλάμε για κάποιον μελλοντικό κανονισμό, θα πρέπει να προστατεύει τη δημόσια υγεία. Δεν θα σχολιάσω λοιπόν ποιος ε, κανονισμός είναι καλύτερος, δεν έχουμε την ε, απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη, αλλά θα πρέπει να φροντίσουμε να ε, προστατευτεί η νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστώ κύριο Κάρανς. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. θα ήθελα να ενισχύσω την αξιοπιστία σας λίγο γιατί λέτε ότι δεν ασχολείστε με τεχνικά θέματα. Και η Επιτροπή μας είναι εν ε, Τεχνική Επιτροπή. Αλλά ποιον εκπροσωπείτε. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Εμείς είμαστε μη κυβερνητική οργάνωση. Δεν έχουμε μέλη, αλλά έχουμε μια σαφέστατη αποστολή η οποία περιγράφεται στην ιστοσελίδα μας. Είμαστε 14 και προσπαθούμε να ερευνήσουμε και να δημοσιεύσουμε στοιχεία για τα λόμπι. Είστε υπέρ της διαφάνειας και της δημοσίευσης όλων των εγγράφων. Ποιος σας χρηματοδοτεί. Στις γραπτές απαντήσεις ε, σας δίνουμε λεπτομέρειες. Έχουμε όλες τις πηγές χρηματοδότησης στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε προϋπολογισμούς για τα έσοδα που έχουμε λάβει τα τελευταία δέκα χρόνια. Και αυτό υπάρχει και στο Μητρό Διαφάνειας. Είστε πολύ ανοιχτοί στην ιστοσελίδα σας αλλά πώς 15 άνθρωποι έχουν δώσει 34%, το 7% όμως, το 4% προέρχεται από ιδρύματα. Είναι το Ίστβαρα, το οποίο χρηματοδότησε το 23% του προϋπολογισμού σας το 15% και 30% τον επόμενο χρόνο. Τι είναι αυτό το Ίδρυμα που χρηματοδοτεί τόσο πολύ, το 1 τρίτο των εργασιών σας. Γιάντε Ιστβάρα είναι ένα Ίδρυμα υποτροφιών, υποστηρίζει τις ΜΚΟ που είναι δραστήριες στον τομέα του περιβάλλοντος και του δημοσίου ελέγχου εφόσον κάθε χρόνο γίνεται το αίτημά μας δεκτό, πράγματι δεχόμαστε μία χρηματοδότηση από πλευράς τους. Τι είναι πίσω από το Ισβάρα. Έχει δημιουργηθεί από ένα φιλάνθρωπο ο οποίος πιστεύει ότι πρέπει να προωθήσει την ενίσχυση των ΜΚΙΟ. Εγώ όταν βλέπω την ιστοσελίδα του Istvara Foundation λένε ότι υποστηρίζει τοπικές εκστρατείες εναντίον των προβληματικών νεοφιλελεύθερων πολιτικών όπως του ΠΟΕ, της Παγκόσμιας Τράπεζας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κτλ. Το Ίστβαρα λέγει ότι είναι ε, μια εκστρατεία ουσιαστικά ε, για την υπονόμευση οργάνων όπως η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ισχύει κάτι τέτοιο. Εγώ δεν το ερμηνεύω με αυτό. Το είναι ένα προοδευτικό ίδρυμα το οποίο ασκεί αξίες προστασίας των κοινωνικών δικαιωμάτων και των οικονομικών δικαιωμάτων δεν είναι θέμα, λέει εδώ, υποστηρίζει τοπικές εκστρατείες εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας υποστηρίζουν για να εκστρατεύετε εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κοιτάξτε, εδώ μιλάμε για συγκεκριμένη, ε, εν περιπτώσει, πολιτική. Και είναι ενδιαφέρον, ε, αλλά το 2015 είχε δημιουργηθεί από τον Άιμαν Τζάλλα, ο οποίος είναι από το Λίβανο, και τα χρήματα προέρχονται από ένα λογαριασμό της UBS. Είναι κάτι σαν τα Panama Papers, είναι μη διαφανής πηγή πληροφόρησης για μια οργάνωση η οποία υποτίθεται προωθεί τη διαφάνεια. Η ερώτησή μας λοιπόν είναι ότι εμείς εδώ ακούμε την κοινωνία των πολιτών και από ό,τι φαίνεται εσείς οι δύο τους οποίους ακούσαμε πριν η κοινωνία των πολιτών σας χρηματοδοτεί κατά 4% και ε, το μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησης προέρχεται από ένα οργανισμό ο οποίος έχει σαν στόχο να καταπολεμήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κοιτάξτε, αυτά είναι θέματα που έχουμε συζητήσει σε επίπεδο δημοκρατικής διαδικασίας με τους συντονιστές. Είναι πολύ δύσκολο να οργανώσει κανείς ε, μια αν θέλετε, αλληλουχία συναντήσεων με αποτελεσματικό τρόπο. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με οργανώσεις οι οποίες ε, είναι εναντίον των νεοφιλελεύθερων ιδεών. Όπως είπα και πριν, εμείς βλέπουμε πάρα πολλές ΜΚΟ, πάρα πολλούς τεχνικούς, και μέχρι τώρα, μην φτάσουμε τη στιγμή αυτή που κάνουμε πολιτικές συζητήσεις, οι ΜΚΟ δίνουν διαφανείς πληροφορίες για τη χρηματοδότησή τους και δεν δικάζονται σήμερα. Ε, σύμφωνο, αλλά αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι μιλάνε για τη διαφάνεια, την ενημέρωση, αλλά σε σχέση με τους εαυτούς τους δεν είναι ιδιαίτερα διαφανείς. Ε, δεν δείχνουν ακριβώς το τι κάνουν. Ίσως και στο γραπτό. Κοιτάξτε, ε, ε, εγώ πρέπει να διευκρινίσω ότι και στις γραπτές απαντήσεις είπαμε ότι είμαστε διαφανείς σε σχέση με τα χρήματα τα οποία λαμβάνουμε. Ο Ίδρυμα Ισβάρα έχει μία δήλωση προθέσεων και αποστολής η οποία είναι συμβατή με τις δικές μας προσπάθειες. Ε, ε, αυτό που είπατε για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ισχύει 100%. Υποστηρίζονται οι ΜΚΟ στον τομέα των ε, περιβαλλοντικό και εναντίον των ε, νεοφιλελεύθερων πολιτικών. Είναι ένα ίδρυμα οργανωμένο με βάση την ελβετική νομοθεσία, έχει λογαριασμό στην Ελβετία ο κύριος Ευχαριστώ πολύ. Εμένα με ενδιαφέρουν περισσότερο οι πληροφορίες που έχετε να μας δώσετε. Το... Νομίζω ότι εμείς θα σχηματίσουμε την άποψή μας για την οργάνωσή σας εν ευθέτω χρόνο. Και ε, η χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν νομίζω ότι εμπίπτει στην ε, εντολή της Επιτροπής μας, αλλά από εκεί πέρα μπορώ να σας ρωτήσω οτιδήποτε. Τι φάγατε για πρωινό και πώς φτάσατε εδώ σήμερα, αλλά θα σας ρωτήσω Σχετικά με τα ευρήματά σας για την βιομηχανία αυτοκινήτων, ε, αναφέρατε ότι έχουν δημιουργηθεί παραθυράκια. Τι αποδείξεις έχετε ή παραδείγματα για αυτά τα παραθυράκια. Ευχαριστώ. Έχουμε τα δεδομένα σχετικά με την μείωση της θερμοκρασίας Ε, άλλαξε το όριο από 0 σε 3 ε, βαθμούς θερμοκρασίας. Ε, Θεωρείται δηλαδή ότι 3 βαθμοί είναι μια μέτρια θερμοκρασία. Επίσης όσον αφορά την, το ξεκίνημα με κρύα μηχανή. σε χαμηλή θερμοκρασία. Και υπήρχε εν μέρη αποδοχή των ε, συνθήκων οδήγησης ε, κατά πόσο ε, γίνεται σε αυτοκινητόδρομο ή στην υπεθροίση της πόλης και η μέγιστη ταχύτητα ε, μειώθηκε από 60 χιλιόμετρα την ώρα. Η πρόταση ήταν στα 130, ε, αλλά τελικά συμβαστήκαμε στα 145, στα 145 χιλιόμετρα την ώρα, ε, αλλά με κατάργηση του τεστ ε, υψηλής ταχύτητας. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε εδώ το ρόλο που έπαιξε η Volkswagen, παρότι ήταν κάτι που κάλυπτε το σύνολο της βιομηχανίας διότι η Volkswagen ε, έστειλε επιστολή στην Γενική Διεύθυνση Grow και της είπε ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν τα όρια ταχύτητας ε, και μην ξεχνάτε ότι η Volkswagen ε, έχει στην κατοχή της ε, και την Porsche και την Lamborghini. Και όταν προσεγγίσαμε την Volkswagen για το θέμα αυτό μας είπε ότι αυτό δεν ήταν lobbying, ήταν κανονική ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης που αποτελεί μέρος της νομοθετικής διαδικασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δεν θα πρέπει να θεωρηθεί lobbying. Και αν έχω το χρόνο θα ήθελα να αναφέρω ακόμα ότι σε εθνικό επίπεδο υπάρχει συντονισμένη προσπάθεια για νέες προτάσεις σε νέα όρια, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα πληρούνται τα, οι προϋποθέσεις της Κομισιόν. Είπατε ότι έχει γίνει ε, εσκεμμένη καθυστέρηση. Μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα. Και όσον αφορά τους ε, παράγοντες συμμόρφωσης που αναφέρατε, μας είπατε ότι χρησιμοποιούνται διάφορες ε, τακτικές. ώστε η βιομηχανία να περάσει ε, τη... αυτά που θέλει η ίδια. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι τακτικές. Έχουμε εδώ πέρα μια διτή προσέγγιση. Πρώτον, να γίνει η ψηφοφορία όσο γίνεται πιο γρήγορα για όλες ε, τις ε, συνθήκες ε, και δεύτερον να προσθεθούν περισσότερες προϋποθέσεις και να καθυστερήσουν τα κριτήρια. κάτι που ήταν πολύ δύσκολο να γίνει εγκαίρως πριν την ψηφοφορία. έτσι λοιπόν ουσιαστικά επρόκειτο για καθυστέρηση της όλης διαδικασίας. Τον Ιούλιο του 2015 υπήρξε ο ισχυρισμό ότι μπορεί να είναι αδύνατο να συμμορφωθεί κανείς με τα κριτήρια και γι' αυτό ζήτησε μια λογική προσέγγιση που απαιτεί ακόμα τεχνικές και πολιτικές συζητήσεις. Και επίσης ε, το έγγραφο που διέρευσε δείχνει ότι τα κράτη-μέλη ε, προσπαθούν να καθυστερήσουν τις διαδικασίες. Επίσης ε, υπήρξαν διάφορες τακτικές, ε, υπήρξε η απειλή για μείωση των ε, θέσεων απασχόλησης. νομικές γνωμοδοτήσεις, συντονισμός των μελών της οργάνωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να γίνονται συντονισμένες επαφές. ώστε να συμπεριληφθούν τα κριτήρια στην ε, διαδικασία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντεμέσμακερ, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε και σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Τώρα, έλαβα τις ε, γραπτές ε, απαντήσεις και τις μελέτησα προσεκτικά και μου κάνει εντύπωση ότι γενικά παραμένετε έτσι πάρα πολύ ασαφείς στις απαντήσεις σας. Και δεν είναι τίποτα που μπορεί να θεωρηθεί έτσι, σκληρή πληροφορία. Σωστά τα λέω. Και μήπως είναι αυτό ένα από τα προβλήματα. Ζητώ συγγνώμη αν θεωρείτε ότι είναι σαφής η απαντήση. Σε ξελίδες είναι. Ε, είναι περισσότερο από οτιδήποτε θα ήθελα να διαβάσουν ε, ε, οι βουλευτές, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ε, περιβάλλοντος ήρθε, έφερε δύο σελίδες και γκρίνιαζαν οι βουλευτές. Ε, παρακαλώ, έχουμε τεχνικές ε, πληροφορίες, έχουμε πολλούς συνδέσμους, ε, αν θέλετε έγγραφα έχουμε να σας φέρουμε και πολύ ε, υλικό. Παρακαλώ, αν στη διάθεσή σας, είναι δημόσια τα έγγραφα, αν θέλετε να τα διαβάσετε, έχουμε πολύ περισσότερη πληροφόρηση, αλλά θεωρήσαμε ότι θα σα ενδιαφέρεται πιο πολύ η ανάλυση και παρά τα έγγραφα. Παρακαλώ, όμως αν θέλετε κάποιες προφορίες είναι στη διάθεσή σας. Η απάντηση στην ερώτηση 4 για παράδειγμα που μιλάτε για ένα έγγραφο το οποίο διέρευσε. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο παραπάνω περί τίνος πρόκειται. Ποιο είναι αυτό ακριβώς το έγγραφο που διέρευσε. So the question for, which is, uh ερώτηση 4 αφορά σε ένα εγγραφό το οποίο δημοσιεύσαμε ε, στην ιστοσελίδα μας. Είναι ένα άρθρο που ε, ε, έχουμε στη διάθεσή σας. Αν δεν το έχουν λάβει τα μέλη να σας το στείλουμε. Είναι ένα στρατηγικό έγγραφο ΑΣΕΑ που λέει τι ε, συμβιβασμοί είχαν γίνει, πώς επηρέασα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ε, τους ελέγχους σε πραγματικό χρόνο, για να υπάρχουν καθυστερήσεις, παραθυράκια και εντάξει. Μάλιστα και στην απάντησή σας υπαριθμών 8 λέτε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει περισσότερη ενημέρωση για τις ομάδες πίεσης, τα λόμπι, η οποία όμως απέχει πόρο από το να είναι ικανοποιητική. Ε, για να ελέγχονται πραγματικά και να παρακολουθούνται τα λόμπι. Λέτε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια, συμφωνώ απολύτως. Αυτό όμως δεν αρκεί ε, για να αποφύγει κανείς την αθέμητη επιρροή. Και στην απάντησή σας στην ερώτηση 12 μιλάτε για τις εδεχόμενες λύσεις για το μέλλον που προτείνετε. Έχω λοιπόν την εξής ερώτηση τώρα. Έχετε παραδείγματα καλών ή βελτίστων πρακτικών σε σχέση με όλα αυτά. Προηγουμένως αναφερθήκατε στην έλλειψη ισορροπίας. σε όλες τις σημαντικές ομάδες οικονομίας ή βιομηχανίας υπάρχουν όμως κάποιοι κλάδοι, κάποιες πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως ε, παράδειγμα προς μίμηση ενδιαφερόμενοι. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας αυτές όσον αφορά τις ε, ομάδες επιρρογνωμόνων και τη σύνθεσή τους. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ομάδων, των οποίων η σύνθεση έχει γίνει πιο ισορροπημένη τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν ε, υπό μεγάλη πίεση. Έχουν λοιπόν γίνει κάποια πολύ συγκεκριμένα βήματα από την Κομισιόν προς την κατεύθυνση αυτή. Ίσως θα είναι χρήσιμο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εσωτερικά να εξετάσει ποιες είναι οι καλύτερες ε, πρακτικές ε, και να τις διευρύνει. Νομίζω ότι αυτό θα ήταν πολύ λογικό. Να χρησιμοποιήσει τις ε, καλύτερες πρακτικές των δικών της διευθύνσεων σε όλες τις διευθύνσεις. Και για περισσότερη διαφάνεια υπάρχουν κάποιες πολύ καλές αρχές σε έγγραφα της Κομισιόν που έχουν να κάνουν με τα νέα πρότυπα διαβουλεύσεων. Θα πρέπει να αποφεύγει να ε, διαβουλεύεται μόνο με τη μία πλευρά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τις ε, επιγραμμικές διαβουλεύσεις, αλλά μπορεί να διευρυνθεί σε όλες τις διαβουλεύσεις της Κομισιόν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Φέντερλεϊ. Βρισκόμαστε σε ένα ε, ευαίσθητο τομέα τα στοιχεία είναι σημαντικά για μας. Δεν μπορούμε να εξαρτώμεθα από ανεξέλεγκτες ε, πληροφορίες. Θα πρέπει να έχουμε δεδομένα πληροφορίες ελεγχόμενες για να λειτουργούμε αποτελεσματικά. Όλοι υφιστάμεθα το λόμπι καθημερινά, μερικές φορές το χρειαζόμαστε αυτό για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε, να κατανοήσουμε και τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις αλλά θα πρέπει αυτό να το διαχειριζόμαστε με τρόπο ελέγξιμο από πλευρά των εκλογέων μας και των ΜΚΟ. Θα ήθελα λοιπόν να δω εδώ αν μπορούμε λίγο να προχωρήσουμε. Η πρώτη ερώτησή μου είναι η εξής. Έχετε κάποιες αποδείξεις ότι έχει υπάρξει σημαντική μορφή επηρεασμού της βιομηχανίας των αποφάσεων που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεύτερη ερώτηση μοιάζει με την προηγούμενη, έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στην ομοθετική διαδικασία. Και τελευταία ερώτηση, αν ναι, και αν έχετε συγκεκριμένα παραδείγματα γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην επαναληφθεί η κατάσταση αυτή, να ακούμε τις απόψεις βέβαια της βιομηχανίας αλλά να τις ελέγχουμε. Ξέρω ότι στις Ηνωμένε Πολιτείες, σαν παράδειγμα, κάποιοι πολιτικοί θέτουν στόχους και αυτό δημοσιεύεται και ασκείται κριτική από τους αντιπάλους και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία τότε λαμβάνονται οι τελικές αποφάσεις. Μήπως αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο θα έπρεπε και εμείς να ακολουθήσουμε. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να δείξουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να δείξουμε ε, ότι υπάρχει άμεση σχέση αιτίας και αποτελέσματο ανάμεσα σε μια συνάντηση και με το σχετικό μαθητικό αποτέλεσμα. Αλλά γνωρίζουμε τις διαδικασίες και βλέπουμε το αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, ε, ότι η διαδικασία δοκιμών ψηφίστηκε το 2015 ε, και το θέμα είναι εάν θα είχαμε καν μια τέτοια πρόταση χωρίς το σκάνδαλο της ε, Volkswagen. Όσον αφορά τους παράγοντες ε, συμμόρφωσης, το 2015 ε, και το 2019 αντίστοιχα για παλιά και νέα αυτοκίνητα θα ισχύσουν οι νέες τιμές. Και βλέπουμε ότι η πρόταση της Επιτροπής ήταν ε, να υπάρχει μία φάση μόνο και βλέπουμε και τα κράτη-μέλη να ασκούν πίεση ε, σύμφωνα, σύμφωνη με την γραμμή της βιομηχανίας αλλά είναι πολύ δύσκολο το θέμα των αποδεικτικών στοιχείων την στιγμή που είναι πολύ περιορισμένη η πρόσβασή μας σε έγγραφα. Έχουμε κάποιες επιστολές, αλλά δεν υπάρχουν πρακτικά των συναντήσεων. Κάποιες από τις συναντήσεις είναι ούτως ή άλλως άτυπες και μόνο λόγω ε, των σκανδάλων και των διαρροών ε, γίνεται κάτι. Δεν έχουμε λοιπόν πλήρη πληροφόρηση. Θα δώσω όμως το λόγο στον συνάδελφό μου όσον αφορά το πώς μπορούμε να αποφύγουμε την ε, υπερβολική επιρροή της βιομηχανίας, νομίζω ότι το αποτέλεσμα που δώσατε ε, σχετικά με την υπηρεσία περιβάλλοντος των ΗΠΑ ε, είναι ενδιαφέρον. Βλέπουμε ότι η βιομηχανία αυτοκινήτων συμμετέχει σε όλη την διαδικασία από την αρχή μέχρι το τέλος και μάλιστα με πολύ έντονο τρόπο. Το θέμα είναι εάν αυτό είναι απαραίτητο και εάν ε, ε, είναι υγιής η διαδικασία αυτή. Μήπως είναι πιο χρήσιμο να έχουμε μία φάση για ε, την θέσπιση των κριτηρίων, μετά έχουμε διαβουλεύσεις ε, και συμβουλές από εμπειρογνώμονες και έτσι αποφεύγεται το lobbying. Ίσως θα ήταν χρήσιμο να σκεφτούμε μια τέτοια διαδικασία. Η προορατική συμμετοχή της βιομηχανίας αυτοκινήτων σε κάθε φάση σημαίνει ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη επιρροή, πόσο μάλλον και με την επιγνωμοσύνη που παρέχει. Θα ήταν χρήσιμο να υπάρχουν κάποιες φάσεις που να έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες και να λαμβάνεται η πολιτική απόφαση χωρίς τη συμμετοχή ε, των ε, λομπιστών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο Δε ε, παρακαλώ. Στα αγγλικά όμω ο κύριο Δε Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και του εκπροσώπου του Observatory Europe. Εδώ δεν σας δικάζουμε. Παρακαλώ ε, καταλάβετε ότι ε, μας βοηθάτε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να καταλάβουμε καλύτερα τη διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Ε, το πρώτο που έχω να ρωτήσω είναι η πρόσβαση στα έγγραφα. Αν δούμε τι ισχύει, έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, Ξέρετε τίποτα για κανόνες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που να λέει ότι έχουν την υποχρέωση να τηρούν πρακτικά και αν όχι το έχετε συζητήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι περίεργο. Ξαφνικά ανακαλύπτουμε νέες συνεδριάσεις που δεν τις γνωρίζαμε και ε, τι ανακαλύπτουν τώρα. Τι μπορεί να γίνει εκεί, τι σα, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεύτερον, εσεί τι σχέδια έχετε σε σχέση με πρόσθετη πληροφόρηση που μπορεί να χρειάζεστε και να ε, μα βοηθήσει και εδώ στην Επιτροπή μα. Απαντήσω στην πρώτη ερώτηση. 13 συνεδριάσεις μας είπανε. Όταν ε, ζητήσαμε πρακτικά μας είπανε ότι δεν είχαν καθόλου πρακτικά καμία από τις 13. Αργότερα το ξαναζητήσαμε μας είπαν ότι έχουν συν 7 συνεδριάσεις και άλλη μία. Α, στις δύο βρήκανε πρακτικά, στις υπόλοιπες όχι. Και μετά δημιούργησαν πρακτικά από προηγούμενες συζητήσεις, ε, από σημειώσεις. Περίεργο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δεν ξέρω αν αφήνεται σε πολιτική πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά το σκάνδαλο Dieselgate και τη διαρροή. Δεν θα προχωρήσω σε εικασίες, αλλά υπάρχουν ε, τις γραμμές και σας διαβάζω, άμα το βρω, τον κώδικα δεοντολογίας. Μια στιγμή που το έχω. Ναι για τις συνεδριάσεις με λόμπι υπάρχει ένας κατάλογος, ένας οδηγός ε, πρακτικός συμπεριφοράς ε, για τη διοντολογία των υπαλλήλων. Στις συνεδριάσεις αυτές θα πρέπει να υπάρχει γραπτή καταγραφή, πρακτικά δηλαδή, σε κάθε περίπτωση που ε, ε, μπορεί να αφορούν δράσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή περιλαμβάνουν σημαντική πληροφόρηση. Αυτά θα πρέπει να πρωτοκολούνται και να αρχιοθετούνται. Δηλαδή φυσικά θα πρέπει και πρακτικά να έχουν και να καταγράφονται αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Αρμόδια Γενική Διεύθυνση Grow δεν το ακολουθεί αυτό και θα θέλαμε να μάθουμε τι μέτρα ελήφθησαν έτσι ώστε στη συγκεκριμένη Γενική Διεύθυνση να καταγράφονται οι συνομιλίες αυτές σε πρακτικά δηλαδή και να τηρείται ο κώδικας. Αλλά από εκεί και πέρα... Δεν ξέρουμε τι βήματα έχει κάνει ε, η ε, για να, για να προστατεύσει τον εαυτό της ε, από σύγκρουση συμφερόντων. Όπως είπε και ο Λιβιέ, υπάρχουν και τέτοιες προβλέψεις. Δεν ξέρω αν έχουν λάβει μέτρα, ασφαλιστικές δικλείδες σε προφυλάξεις, έτσι ώστε η πολιτική διαδικασία λήψη των αποφάσεων να προστατεύεται από την επιρροή τέτοιων συμφερόντων και από τη σύγκρουση συμφερόντων. Να προσθέσω και άλλο ένα θέμα, διότι μας τελειώνει ο χρόνος συστήνεται όλες οι επαφές προσωπικού της Κομισιόν με λομπίστες να καταχωρούνται και να δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα, όπως ισχύει ε, και για τους ε, επιτρόπους και τους γενικούς διευθυντές. Ρώτησα όμως ε, και μου είπαν ότι αυτό μπορεί να είναι παραβίαση του ιδιωτικού βίου των εμπλεκομένων. Ποια είναι η θέση σας γι' αυτό. Και όσον αφορά τις άτυπες ε, συναντήσεις εκτός ε, της, ε, εκτός της Κομισιόν, σε ξενοδοχεία ή σε άλλα μέρη, πώς, θεωρούνται, πώς τις αντιμετωπίζουμε, θεωρούνται συναντήσεις? Πιστεύουμε ότι η διαφάνεια στις συναντήσεις με τα λόμπι είναι βασική. Αυτό θα επιτρέψει καλύτερο έλεγχο των επαφών και των συνεννοήσεων ανάμεσα στους λόμπι και τις αρχές. Η ανησυχία για την ιδιωτικότητα ή την εμπιστευτικότητα είναι κάτι το θεμητό. Νομίζω ότι τα ονόματα των κατώτερων ας πούμε ιεραρχικά υπαλλήλων μπορεί να μην περιλαμβάνονται αλλά η, υπηρεσία και το όνομα του υπεύθυνου μιας υπηρεσίας νομίζω είναι κάτι το οποίο θα ήταν επαρκές σε επίπεδο ενημέρωσης. Το σημαντικό είναι ότι οι συναντήσεις έγιναν σε όλα τα επίπεδα και ε, είναι σημαντικό τμήμα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και γι' αυτό θα πρέπει να δημοσιοποιούνται, να είναι διαθέσιμες προς έλεγχο. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Λέει η κυρία Ντέλη, όταν μιλάμε για τα λόμπι αυτό ακούγεται ύποπτο, αλλά τουλάχιστον το συζητάμε. Να έλθω στην απάντηση που δώσατε στην 10. Πέρα από τη διαφάνεια πρέπει να στείλουμε στους ευρωϊπαλλήλους, στους υπεύθυνους ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις επαφές τους με τα λόμπι. Πρέπει να υπάρξει πολλαπλότητα εμπειρογνωμοσύνης και πλήρης ανεξαρτησία από τον τομέα ο οποίος είναι το αντικείμενο της μελέτης. Ε, μια ειδική ομάδα λοιπόν η οποία ήταν ε, με βασικό στόχο το Euro 5, Euro 6 υπήρχαν ε, εκπρόσωποι των εταιριών και από την άλλη υπήρχε και η Ομοσπονδία η Παγκόσμια Αυτοκίνητο Παραγωγής και υπήρχε μόνο ένα, μία μικιό περιβαλλοντική. Πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να θεωρούνται οι κατασκευαστές σε σχέση με το Euro 5 και Euro 6 ε, συνομοθέτες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ΚΑΣ 21 λοιπόν η συγκεκριμένη αυτή συνάντηση ήταν μια εξαιρετική πρωτοβουλία από τον τότε Επίτροπο Φερχόιγκεν για την δημιουργία μιας ομάδας υψηλού επίπεδου η οποία ήταν ακραία μη ισόρροπη είναι ένα από τα χειρότερα παραδείγματα τα οποία μπορεί να βρει κανείς στην ιστορία αυτών των επαφών. Είχαμε τους προέδρους των Δημοκητικών Συμβουλίων των μεγάλων Αυτοκίνητων Βιομηχανιών και υπήρχε μία μόνη ε, περιβαλλοντική. Ασκήθηκε κριτική και τότε και όταν ξεκίνησε ξανά η ομάδα μετά από λίγα χρόνια υπήρξε μια καλύτερη ισορροπία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε το μήνυμα αν θέλετε ότι τα αιτήματα των λόμπιστ από πλευράς της αυτοκινητοβιομηχανίας θα πρέπει να αντιπαρατίθενται και με άλλη εμπειρογνωμοσύνη και απόψεις. Υπήρξε παραγωγή πολλών εκθέσεων από, την, από αυτό το επίπεδο επαφών, το κάσι το για την βιομηχανία ο στόχος ήταν να προτείνουν τις δικές τους απόψεις βέβαια για την σωστότερη και ορθότερη νομοθετική ρύθμιση η οποία να ήταν πιο ήπια θα έλεγα να μην φύγει τις αυτοκίνητο-βιομηχανίες να προωθεί την από ρύθμιση και αυτορύθμιση επίσης. Μετά από τις πρώτες εκθέσεις ήταν ικανοποιημένες οι βιομηχανίες από το περιεχόμενό τους, θεώρησαν ότι ήταν συμβατές με τα συμφέροντά τους και τις αρχές τις οποίες είχαν ε, ε, συμφωνήσει, με τις οποίες είχαν συμφωνήσει. και ήταν πολύ σημαντικό επιτροπές όπως η δική σας να αξιολογήσουν ε, τέτοιου είδους διαδικασίες. Νομίζω ότι στην ουσία έχουν αλλάξει κάπως τα πράγματα από τότε. Ευχαριστώ. Εγώ βλέπω τα πρακτικά της ομάδας αυτής του ΚΑΣ 21. Υπάρχει ανάγκη να εξετάσουμε το Euro 5 και Euro 6 υπό το φως της ορθότερης νομοθετικής ρύθμισης, κάτι το οποίο επιτρέπει περαιτέρω αυτορύθμιση αυτή η ομάδα, το ΚΑΡΙ 21, ε, μήπως ήταν ένα μέσο αυτορύθμισης των αυτοκίνητων βιομηχανιών στα πλαίσια και εξ ονόματος της καλύτερης νομοθετικής ρύθμισης. Μαζί με τους φίλους της Γης ε, εμείς θα δημοσιεύσουμε το Σεπτέμβριο μία έκθεση, θα την υποβάλουμε και στην Επιτροπή σας. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, δεν μπορούμε να δώσουμε μια πλήρη απάντηση ε, υποτίθεται ότι και το EU Observer θα κάνει μία έρευνα σε σχέση με τέτοιου είδους πρακτικές. Πράγματι το ΚΑΒΣ 21 υιοθέτησε τις απόψεις της βιομηχανίας, ιδιαίτερα τους αυτοελέγχους όπως λέγονται και τις δοκιμές τις οργανωμένες από τις ίδιες τις βιομηχανίες και χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθούν πολλοί τομείς βιομηχανικής δραστηριότητας. Νομίζω ότι είναι κάτι το πολύ συγκεκριμένο και κάτι το οποίο θα πρέπει με ε, πολύ προσοχή να εξεταστεί εκ νέου. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Εύη, για την προσπάθεια την οποία κάνετε μέχρι τώρα και για τις πληροφορίες τις οποίες μας δώσατε σε πάρα πολλούς τομείς Σκέφτομαι επίσης και το θέμα των διαταρακτών, των ενδοκρινικών ε, διαταρακτών. Έχετε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σαν οργάνωση και σας ευχαριστώ που συμμετέχετε και στην σημερινή μας συνάντηση. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό όταν ομιλώ σαν πολίτης Ευρωπαίος να γνωρίζω ότι πέρα από τις επαφές οι οποίες γίνονται κατά κάποιο τρόπο σε τακτικό επίπεδο στο εσωτερικό των ευρωπαϊκών οργάνων με σαν παράδειγμα με στόχο ας πούμε το Μητρό Διαφάνειας έτσι ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορέσει να ξεπεράσει τα όρια τα οποία έχει λειτουργία σε σχέση με τον τομέα αυτό. Υπάρχει όμως κάτι που με ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Είναι η παρουσία επαφών με τον βιομηχανικό κόσμο σε επίπεδο τεχνικό. Γιατί όπως και εσείς μας είπατε είναι πάρα πολύ συχνό ε, η, συνεργασία, η συνεισφορά της βιομηχανίας στην ουσία μερικές φορές καλύπτεται πίσω από τη μάσχα της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης που λείπει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε κάποιες προτάσεις για να λυθεί το θέμα αυτό. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων εσείς πιστεύετε ότι τα ευρωπαϊκά όργανα είναι δεκτικά, είναι ε, ανοιχτά στο να δεχθούν κάποια από τα μέτρα τα οποία εσείς έχετε προτείνει έτσι ώστε να βελτιωθεί η σχέση με τον βιομηχανικό κόσμο ή εξακολουθούν να είναι απόλυτα μη δεκτικοί. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το Μητρό Διαφάνειας, αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα πρόοδου, αλλά υπό τη μορφή που έχει αυτή τη στιγμή δεν έχει την αξία που θα μπορούσε να έχει. Ε, εντός του έτους ε, ο πρόεδρος Γιούγκερ υποσχέθηκε ότι θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες για ένα νέο μητρό. Ελπίζουμε ότι θα γίνει υποχρεωτικό αυτό. Δεν διασφαλίζει όλοι οι λομπίστες να το υπογράφουν και να υποβάλουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Ε, σημαντικό είναι να διασφαλιστεί η αξιοπιστία των πληροφοριών και η ε, ε, επικαιροποίηση των πληροφοριών, διότι πολλές πληροφορίες που υπάρχουν στο Μητρό Διαφάνειας δεν έχουν ελεγχθεί και δεν είναι αξιόπιστες και επικαιροποιημένες. Ελπίζουμε λοιπόν η αναθεώρηση αυτή που θα ξεκινήσει το φθινόπωρο να βελτιώσει τα πράγματα ώστε να έχουμε πρόσβαση σε επίκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες. Η δεύτερη ερώτηση είχε να κάνει με τις επαφές ανάμεσα στους νομοθέτες ή τους αξιωματούχους της Κομισιόν και την, και την σχετική βιομηχανία. Χρειαζόμαστε μια πιο επίσημη προσέγγιση και να υπάρχει η δυνατότητα να προστατεύονται οι υπάλληλοι της Κομισιόν από την πίεση από πλευράς ε, της βιομηχανίας. Αυτό πρότεινα και πριν, ε, μιλώντας για ένα time out, μια φάση στην νομοθετική διαδικασία όπου να μην ε, συμμετέχουν οι λομπίστες. Εφόσον δηλαδή έχουν συγκεντρωθεί όλες οι πληροφορίες, έχει γίνει η διαβούλευση, να υπάρχει χρόνος ε, για τους ε, αξιωματούχους της Κομισιόν να πάρουν το χρόνο τους ε, μακριά από την επιρροή άλλων. Στα τέλη του 2013, αρχές του 2014, ο τότε Επίτροπος Μπαρνιέ αποφάσισε να υπάρξει τρίμηνη πάυση συναντήσεων με λομπίστες για ένα συγκεκριμένο θέμα διότι θεωρούσε ότι οι υπάλληλοι του χρειάζονται το χρόνο να συγκεντρωθούν για να εκπονήσουν την καλύτερη δυνατή πρόταση. Έτσι λοιπόν ε, για μια τρίμηνη πάυση επαφών. Αυτό νομίζω θα ήταν χρήσιμο να γίνεται. Ωραία, σας ευχαριστώ. Ε, έτσι ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Προχωρούμε στο δεύτερο γύρο. Δίνω το λόγο στην κυρία Τούνου Αινστάιν. Ευχαριστώ πολύ. Μιλάμε πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πάντως για τις πληροφορίες σας, για τις πρακτικές, για τη διαφάνεια και τα λοιπά. Θα ήθελα όμως να έρθω στην νομοθετική διαδικασία και σε σχέση με τις ε, εκπομπές NOx. Εσείς βλέπετε ότι Υπάρχουν προβλήματα στις προσπάθειες τις οποίες έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αν ναι, ε, ποια είναι αυτά τα προβλήματα. Σίγουρα υπάρχουν αδυναμίες. Εμείς σαν οργάνωση συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά αυτό είναι πρόβλημα και σε διεθνές επίπεδο πρέπει να υπογραμμίσω την εμπλοκή και την εξάρτηση από την εμπειρογνωμοσύνη της αυτοκινητοβιομηχανίας που οδήγησε σε ρυθμίσεις σε σχέση με τα νόξ και τα κόξ τα οποία στην ουσία θα έλεγα ευνοούν τα συμφέροντα των οικονομικών εμπλεκομένων εταίρων. Η εμπειρογνωμοσύνη που θα έπρεπε να υπάρχει στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το πώς θα μονώσουμε την ομοθετική διαδικασία εδώ υπάρχουν προτάσεις εφόσον σας ενδιαφέρουν. Πάντως υπάρχουν ε, ε, προβλήματα και σε τεχνικό και σε πολιτικό επίπεδο. Το πώς ε, βασίζεται στην εμπειρογνωμοσύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν δεν την έχει είναι θέμα που έχει και πολιτικές αν θέλετε διαστάσεις. Η επιλογή του από πού θα προέλθει η εμπειρογνωμοσύνη που ελείπει εσωτερικά είναι μια πολιτική επιλογή. Πρέπει λοιπόν να σταλεί ένα πολιτικό μήνυμα το οποίο να λέγει ότι η εμπειρογνωμοσύνη αυτή θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη πραγματικά. Έχετε τεχνικές ε, προτάσεις συγκεκριμένες. Κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε μέρος στις ομάδες εμπειρογνωμόνων. Ε, η ομάδα εμπειρογνωμόνων για το RDE. Ε, υπάρχει ανάγκη φυσικά για την τεχνογνωσία της βιομηχανίας. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε εδώ μας δίνουν σωστά παραδείγματα σε σχέση με τη συνεργασία τους με το Διεθνές Ινστιτούτο ε, πρόληψης του καρκίνου. Υπήρξαν ε, ομάδες εργασίας σε δύο επίπεδα. Στη μία υπήρξε ε, μια ομάδα εργασίας με αυτούς που δεν είχαν οικονομική εμπλοκή και στο δεύτερο επίπεδο αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται οικονομικά και είχαν συμφέροντα σε σχέση με την τελική νομοθετική πρόταση. Η πρώτη ομάδα η δεύτερη ομάδα μάλλον καλείται από αυτούς, συγκαλείται από την πρώτη ομάδα σύνα τμήματα της δεύτερης όταν αυτή θεωρείται απαραίτητη και όταν θεωρείται ότι τα συμφέροντά τους δεν θίγονται. Η κυρία Ρεβό. Μετά από τις απαντήσεις που δώσατε στο ερωτηματολόγιο φαίνεται ότι η κακοδιαχείριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυταπόδεικτη. Ελλείψεις γνώσης, έλλειψη διαφάνειας, μη απαντήσεις κτλ. κτλ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι σκοπούμενο ή μη. Υπάρχει τρόπος ε, να πάρουμε μια απόφαση που να αλλάξει επιτέλους αυτή η κατάσταση. Δεν είναι δυνατόν για μας να κρίνουμε αν τα προβλήματα αυτά είναι, έγιναν επί τούτου, προκλήθηκαν επί τούτου ή αν υπάρχει μια αδυναμία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν είναι έτοιμη να προχωρήσει στις σωστές διαδικασίες ελέγχου. Ο οδηγός διοντολογίας δεν εφαρμόζεται ιδιαίτερα από την Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης από ό,τι φαίνεται έχουν δημιουργηθεί κάποια έθιμα στο εσωτερικό αυτού του τμήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία δεν σέβονται τη διαφάνεια και δεν σέβονται τις προσπάθειες προστασίας των διαδικασιών λήψης απόφασης από εξωτερικές παρεμβάσεις. Στην απάντησή σας ερώτηση 4 Όντω και εγώ χρειαζόμουν περισσότερε λεπτομέρειε, Αρχίσατε κάπως να απαντάτε και έχει αρκετό ενδιαφέρον. Η επιρροή λοιπόν το, της βιομηχανίας οδήγησε σε αλλαγή κάποιων στοιχείων όπως είναι οι θερμοκρασίες, ε, κάποιες άλλες δοκιμές ε, εξαιρέθηκαν. Θα μπορούσατε γραπτός να μας απαντήσετε εδώ, μας δώσετε παραδείγματα και από ό,τι φαίνεται έχετε κι άλλα. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο για μας να έχουμε και τα υπόλοιπα πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Κατά τα άλλα γίνεται μέγας λόγος για τη Volkswagen. Οι άλλοι κατασκευαστές τι έκαναν. Συμμετείχαν, επηρέασαν τα πράγματα τις τελευταίες ε, αποφάσεις ε, του CTVM σε ό,τι αφορά για την επιρροή για τις συγκεκριμένε δοκιμές. Εμείς τι κάναμε. Ε, συγκρίναμε τα αρχικά έγγραφα με το τελικό ε, αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έγινε το α που είχε τη συγκεκριμένη επίπτωση, αλλά ε, κάποια πράγματα βγήκαν, αποδυναμώθηκε το κείμενο για όρια ταχύτητας, για ταχύτητες, για... Ε, υπάρχει μια ολόκληρη λίστα συνθήκες οδήγησης, αν θέλετε μπορώ να σας δώσω τον πλήρη κατάλογο. Επίσης, θα έρθει και άλλο πακέτο για τις δοκιμές σε συνθήκες πραγματικής οδήγησης. Δικό σας θέμα είναι αυτό. Εγώ είμαι από την κοινωνία των πολιτών. Τώρα η επιρροή αν είναι από την αυτοκινητοβιομηχανία που θέλει να τα ξεφορτωθεί, δεν ξέρω. Δεν είναι καθόλου πρόβλημα ο Volkswagen, είναι πρόβλημα αυτοκινητοβιομηχανίας και από τη Ford υπάρχει μεγάλη πίεση, από την BMW, Daimler. Ε, το έγγραφο όμως που διέρευσε μπαίνει σε λεπτομέρειες για το ποιος ηγείται η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία στατή. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τους Γερμανούς και είναι και συντονισμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το σύνολο της αυτοκινητοβιομηχανίας, δεν είναι κάποιος τυχαίος που ήρθε κάτι να πιέσει. Ο κύριος ε, Σούλτζαν. Ε, και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να συζητήσουμε. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να επανέλθω στην παρουσίαση με PowerPoint της ΑΣΕΑ που στις 16 Μαρτίου αφήσατε να διαρρεύσει και ο Πολ Γουίνιγκ από την ΑΣΕΑ συζήτησε λέτε με τον κύριο Στάινιγκερ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Στάινιγκερ δεν είναι γνωστός ως λόμπι αυτοκινητοβιομηχανίας, ε, φιλικός. Είναι πάρα πολύ αντικειμενικός υπάλληλο και τουλάχιστον εγώ έτσι το αξιολογώ. Και με μια τέτοια δημοσίευση κινδυνεύει να μαυρωθεί η εικόνα του και να έχει συνέπειες για τον υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, μπορεί να τον ε, μετατάξουν, να τον μεταθέσουν, να τον αθέσουν άλλο χαρτοφυλάκι κτλ. Αυτό για σας είναι ανετική επίδραση μια τέτοια δημοσίευση ή όχι. Ειδικά για εκείνους που κάνουν τη δουλειά τους που θεωρούν ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχουν υπάλληλοι ε, που πρόσκειται στην Αυτό Όταν ένας τόσο σημαντικός ε, υπάλληλο μετατίθεται, αυτό είναι καλό ή κακό. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Νομίζω ότι το έγγραφο που διέρευσε δείχνει ότι υπήρξε συνάντηση σχετικά με τις εκπομπές ε, στην ΑΣΕΑ, αλλά το θέμα αυτό δεν είναι πρωτοβουλία ενός ανθρώπου. Είναι πολύ ευρύτερο πρόβλημα εντός της Γενικής Διεύθυνσης ε, για την Ανάπτυξη. Η όλη σχέση με την ΑΣΕΑ ε, που επιτρέπει μια τέτοια άτυπη συνάντηση. Εξετάσαμε όμως την κατάσταση, δεν έχει χάσει τη δουλειά του αυτό ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ε, καμία πειθαρχή διαδικασία. Έπρεπε να δημοσιεύσουμε εμείς το έγγραφο αυτό, γι' αυτό ήταν απαραίτητο να δημοσιεύσουμε το όνομά του. Δεν είναι όμως προσωπικό το θέμα, είναι πολύ ευρύτερο και δείχνει την εξουσία της βιομηχανίας αυτοκινήτων, την στενή της σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το πώς ε, τα κράτη-μέλη ε, χρησιμοποιούν την ε, επιρροή τους. Μήπως έχω χρόνο για άλλη μια σύντομη ερώτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην απάντησή σας στην ερώτηση 3. Είμαι μηχανολόγος, δεν γνωρίζω πολύ καλά. Μηχανικός. Μηχανικός, δεν μιλώ πολύ καλά αγγλικά. Τι είναι ο προοδευτικό φιλάνθρωπο που αναφέρεται εδώ. Φιλάνθρωπος ε, ε, ε, είναι ένας πλούσιος άνθρωπος με ιδανικά που θέλει να υποστηρίξει καλές προσπάθειες στην κοινωνία, σύμφωνα με τη γνώμη του. Και γι' αυτό δημιουργεί ένα ίδρυμα που κάνει χορηγίες. Αυτό μπορεί να το κάνει κάποιος μόνος του ή μια ομάδα μελών μιας οικογένειας, ε, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Ο κύριος Έρτοχ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά, καλωσορίσατε και από πλευρά μου. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ και χαίρομαι που υπάρχετε γενικώ. Ε, και πολύ καλά που έρχεστε να σταθείτε απέναντι στον ασίδωτο και το νέο φιλελευθερισμό και το γεγονός ότι η δεξιά εδώ σας επιτίθεται και προσπαθεί να υπονομεύσει την ακεραιότητά σας, μη σας πειράζει, έτσι τα συνηθίζουν αυτοί. Ε, πρόσφατα είχαμε μια ενδιαφέρουσα ακρόαση με το λεγόμενο Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η εκπρόσωπος του κέντρου, ανάλογα όπως τη βόλευε, παρουσίαζε το κέντρο της είτε ως ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο, είτε ως ε, ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξαρτάται απολύτως από τις δικές της εντολές. Εσείς ξέρετε να έχει επιρροή άμεση ή έμεση καμιά ομάδα βιομηχανίας λόμπι ε, στο κοινό κέντρο ερευνών και το θεωρείτε πιθανό να μην είναι πια και τόσο ανεξάρτητο το κέντρο αυτό όπως ισχυρίζεται το ίδιο. Μάλιστα. Στα έγγραφα που λάβαμε εμφανίζεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών γιατί συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία και μια ομάδα task force για τις νέες ε, ρυθμίσεις. Ε, δεν ξέρω. Συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και με τη βιομηχανία το ότι εξαρτάται η εντολή της από την ε, ε, βιομηχανία, όταν κάναν για την υδρορογμάτωση μια έρευνα, το 70% των εκπροσώπων ήταν από τον κλάδο αυτό. Το θέμα είναι ε, ποιος χρηματοδοτεί αυτά. Ε, δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται από τη βιομηχανία, αλλά έχει να κάνει με την πολιτική εντολή που λαμβάνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάστοτε ε, το Κοινό Κέντρο Ερευνών και πώς χρησιμοποιούν τις πληροφορίες με πολιτικό τρόπο. Ε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Ε, ε, θέλουμε να το δούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Προς το παρόν δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω. Θα σας στείλουμε τα στοιχεία. Ευχαριστώ κύριε Σερτούκ. Έχω και άλλη ερώτηση. Τώρα ε, έχουμε την ε, ανανέωση της οδηγίας, μάλλον του κανονισμού για την έγκριση του τύπου, δηλαδή με ποιους κανόνες εγκρίνονται τα νέα μοντέλα για να κυκλοφορούν στην αγορά. Αυτή τη ε, συζήτηση θα την παρακολουθείτε κι εσείς. Πώς θα πρέπει να γίνεται η έγκριση τύπου και να παρακολουθείτε η αγορά για να κλείσουν τα περίφημα παραθυράκια και αβεβαιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι στο οποίο θα ευχαστούμε, να, θα ξεκινήσουμε να εξετάζουμε σύντομα, ιδιαίτερα σε εθνικό επίπεδο. Είμαστε σε επαφή με άλλες οργανώσεις οι οποίες ε, εργάζονται ήδη στον τομέα αυτό. Θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς διαδικασίες, σαν παράδειγμα, ακολουθούνται για τις εγκρίσεις τύπου σε εθνικό επίπεδο. Είναι κάτι το οποίο δεν θα αντιμετωπιστεί μόνο σε επίπεδο επιτροπής ή μόνο σε επίπεδο εθνικών κυβερνήσεων. Τα μαθήματα τα οποία έχουμε πάρει από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επίπεδο διαφάνειας θα πρέπει να εφαρμοστούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών μελών υπεύθυνε για τις εγκρίσεις τύπου. Και κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμβαίνει. Χένκελ. Uh, Αναφερθήκατε επανειλημμένα στον μεγάλο αριθμό των συναντήσεων με λόμπιστα από την αυτοκίνητο βιομηχανία. Η αυτοκίνητο βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη ε, βιομηχανία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ε, έχουμε πάντα μια ηγετική θέση γιατί εκπλήσει λοιπόν το ότι υπάρχουν τόσες πολλές συναντήσεις. Ε, ξέρουμε ε, αντίστοιχα στοιχεία για την υφαντουργία σαν παράδειγμα. Πράγματι είναι το 4% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Ε, το θέμα είναι ότι συγκεντρώνεται σε πάρα πολύ λίγα χέρια. Θα δείτε ότι ο αριθμός των παικτών είναι πάρα πολύ μικρός. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Δεν εκπλήσει λοιπόν το ότι υπάρχουν βιομηχανίες με την αυτοκίνητο βιομηχανία. Λοιπόν υπάρχουν πολλές συναντήσεις και αυτό δεν εκπλήσει. Το επίπεδο όμως πρόσβασης που έχουν στα πλαίσια της διαδικασίας ε, της νομοθετικής, η συμμετοχή τους στην επιτροπολογία κτλ. είναι αυτό το οποίο εκπλήσει. Ε, το θέμα είναι ε, πώς θα στηρίξουμε την αυτοκινητοβιομηχανία χωρίς να ε, υπονομεύσουμε άλλα συμφέροντα της Ένωσης. Εσείς αναφέρεστε σε μορφές συνεργασίας στις μεγάλες επιχειρήσεις μάλλον. Οι λόμπιστ αυτοί ανήκουν στις μεγάλες βιομηχανίες στις ομοσπονδίες, στις εθνικές, εξετάζεται λίγο και τις οργανώσεις των λόμπιστ. Όλοι όσοι εμπλέκονται στις διαδικασίες επηρεασμού των διαδικασιών λήψης απόφασης πρέπει να θεωρούνται λόμπιστ. Εμείς λοιπόν παίρνουμε στοιχεία από το Μητρό Διαφάνεια στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και μια τελική ερώτηση. τα τελικά συμπεράσματα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί από πλευρά της αυτοκινητοβιομηχανία που συναντούν πάρα πολύ συχνά τους εκπροσώπους της Επιτροπής. Μήπως να κάναμε κριτική και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το ότι δεν δείχνει τον ίδιο ζήλο σε ε, οργανωμένα λόμπι ας πούμε του τομέα του περιβάλλοντος ή κάποιων άλλων τομέων. Κοιτάξτε υπάρχει μια τεράστια διαφορά πόρων. Η Volkswagen το 2014 είχε ξεκαθαρά κέρδη που ξεπερνούσαν τα 10 δις. Νομίζω ότι ο προϋπολογισμός της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής της συγκεκριμένη Γενικής Διεύθυνσης δεν ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Υπάρχει μια τρομακτική ανισότητα. Το θέμα δεν είναι να το ισορροπήσουμε αυτό προσκαλώντας περισσότερους εκπροσώπους. Το θέμα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συλλέξει ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και επαϊωσύνη για να μπορέσει να εξισορροπήσει τις σχέσεις της με την αυτοκινητοβιομηχανία. Το θέμα είναι να έχει τις γνώσεις που απαιτούνται. Ο κύριος Ντάνς. Σχετικά με την επιτροπολογία. Είπατε ότι πρέπει να τεθεί το θέμα ακριβώ και των εθνικών εμπειρογνωμόνων που συμμετέχουν σε αυτή. Γνωρίζουμε για αυτούς τι πιστεύετε εσείς ότι είναι ο ρόλος τους, πώς μπορεί να βελτιωθεί η συμμετοχή τους. Εσείς θέλετε να προωθηθεί η διαφάνεια. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε έτσι ώστε οι αποφάσεις να είναι διαφανείς και ταυτόχρονα να δημοσιοποιούνται. Η επιτροπολογία προεδρεύεται είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από τα κράτη-μέλη είναι ένα μαύρο κουτί, δεν ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα εκεί. Έχουμε λίγα έγγραφα και είναι κάτι το οποίο δημιουργεί πολλά προβλήματα και μεγάλη σύγχυση στις Βρυξέλλες. Πρέπει να επαναξεταστεί λίγο η διαδικασία αυτή γιατί ήδη στη συγκεκριμένη περίπτωση του RDE η διαδικασία που ακολουθείται θα επηρεάσει ιδιαίτερα. Κάναμε μία μελέτη λοιπόν για το λόμπι των αυτοκίνητων βιομηχανιών εδώ στις Βρυξέλλες η, ε, ε, η βιομηχανία αυτή στηρίζει τα μέλη του προσωπικού έτσι ώστε της Επιτροπής για να έχουν την πλήρη ε, γνώση τη οποία απαιτείται για τη σωστή του συμμετοχή. Απαιτείται λοιπόν μεγαλύτερη διαφάνεια και αν δεν έχουμε αυτή τη διαφάνεια είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουμε να κάνουμε τον έλεγχο που απαιτείται απαιτούνται κανόνες για ανεξαρτησία και δεύτερον απαιτούνται ε, στοιχεία διαφάνειας. Πιστεύετε ότι υπάρχει μια χώρα η οποία ασχολείται ε, με την αυτοκινητοβιομηχανία περισσότερο από άλλες και σε ποιο βαθμό επηρεάζει αυτό τον τρόπο λειτουργίας. Εμείς δεν είμαστε ούτε στο TCNV ούτε στο RDE. Βλέποντας τα έγγραφα όμως μετά από το διαρρεύσαν μάλιστα έγγραφο βλέπουμε ότι και ποια είναι τα σχόλια που έγιναν για τη διαδικασία της Επιτροπής αντικατοπτρίζονται τα σχόλια ε, και στις ε, απόψεις χωρών όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ιταλία σε σχέση κυρίως με τους παράγοντες συμβατότητας ή συμμόρφωσης δεν ήθελαν κάτι τέτοιο, δεν ήθελαν αυτά τα ποσοστά το 300% για το 2015. Η Ισπανία επίσης είναι παραδοσιακά εμπόδιο. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο και σε εθνικό επίπεδο να υπάρχει διαφάνεια, γιατί πάρα πολύ συχνά πηγαίνουν οι κυβερνήσεις στις πρωτεύουσές τους και κατηγορούν τις Βρυξέλλες, κάτι το οποίο το επιτρέπει δυστυχώς το σκοτεινό, ε, αν θέλετε, χρώμα των διαδικασιών επιτροπολογίας. Ευχαριστώ. Η συνάδελφος προηγουμένως έκανε μια συγκεκριμένη ερώτηση, λέει ο κύριος Σαλίνη. Θα την αναδιατυπώσω εκ νέου. Είναι σαφής ο στόχος της οργάνωσής σας και προσπαθούμε να το συνδυάσουμε με τον δικό μας στόχο για το αν θα πρέπει να ασκηθεί κριτική στα ακράτη μελη και στα ευρωπαϊκά όργανα. Το αίτημα. Εσείς εντοπίσατε συγκεκριμένα προβλήματα στο διακανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των ευρωπαϊκών οργάνων γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, το θέμα των εκπομπών. Έχετε λοιπόν βρει συγκεκριμένα προβλήματα, αδυναμίες σε σχέση με το τι κάνουν τα κράτη-μέλη για τον έλεγχο της αγοράς και τον έλεγχο της εκπομπής καυσαερίων. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε συγκεκριμένα θέματα αν υπάρχουν, όχι το πώς δημιουργούνται τα προβλήματα, αλλά ποια είναι. Όταν υπάρχουν προβλήματα έλλειψης διαφάνειας κτλ. Και φέτο και το τελευταίο κομμάτι της ερώτησής μου για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Αν εσείς έχετε υπόψη σας κάποιες απατηλές παράνομες από πλευράς αυτοκίνητο-βιομηχανιών που έχουν σαν στόχο το να παραπλανήσουν τα αποτελέσματα σε σχέση με τα αποτελέσματα των ελέγχων μετά το 2015 όταν ήρθε σε επιφάνεια η γνωστή ε, περίπτωση της χρήσης λογισμικού που δεν επέτρεπε τη σωστή καταγραφή. Θα πρέπει και πάλι να τονίσω ότι δεν είμαστε οργανισμός που κάνει τις δοκιμές. Δεν έχουμε σχέση με τις δοκιμές εμείς. Μια συμπληρωματική. Καταλαβαίνω αυτή την αντίδραση όταν μετά από όλες τις απαντήσεις που λέτε ότι εμείς δεν απαντούμε επί την ουσία ε, ε, έρχονται κάποιες ερωτήσεις αναπόφευκτες για τη φύση της οργάνωσής σας και όταν ε, είναι προβληματικές οι απαντήσεις σε σχέση με τις δύσκολες αυτές ερωτήσεις είναι δύσκολο να υπάρξει διάλογος. Γι' αυτό απαντήστε επί της ουσίας. Την πρώτη ερώτηση σας απάντησα, έδωσα ε, απαντήσεις, θα υπάρξουν και γραπτές, υπάρχουν δημοσιεύματα, άρθρα. Μπορείτε να δείτε ακριβώς ποια είναι τα παραθυράκια. Συγγνώμη που δεν απαντώ τώρα, θα σας στείλουμε γραπτές απαντήσεις. Ε, όταν υπάρχουν συσκευές εξαπάτησης, πώς καλύπτεις από αποκαλύπτεις την απάτη. Πρέπει να κάνει δοκιμές. Εμείς οργανισμό δοκιμών δεν είμαστε. Δεν πάει ένα μηχανισμό να τα ψάξει δικό μα, αυτά, ή ένας μηχανικός μάλλον. Ε, εμείς ασχολούμαστε με τα λόμπι, με τις ομάδες πίεση. Εμείς θέλουμε να δούμε θεσμικά πώς επηρεάζει ε, η αυτοκινητοβιομηχανία τις ε, αποφάσεις όταν δεν πληρούν τα κριτήρια για τον κινητήρα Euro 6. Εμείς δεν μπαίνουμε σε επιστημονικές λεπτομέρειες και τεχνικές. δυστυχώ, δεν έχουμε τέτοια εντολή. Ο κύριος Γκίζικε. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Σαββίδο και κύριε Χούντεμαν. Εγώ θέλω να επανέλθω στις γραπτές σας απαντήσεις σε ερωτήσεις μας και εσείς επικρίνετε την υπερβολική επιρροή ε, των ε, εκπροσώπων της αυτοκινητοβιομηχανίας σε νομοθέτες και εκπροσώπους της Βρυξέλλης και με στοιχεία προσπαθείτε να το στοιχειοθετήσετε και λέτε ότι κάνουν τις περισσότερες ε, δαπάνες για λόμπι στις Βρυξέλλες και έχουν πάνω από 100 λόμπιστ 5 εταιρείε που τουλάχιστον ένα δακλάσμα του χρόνου τους το αφιερώνουν στο να επηρεάζουν την πολιτική στις Βρυξέλλες. Εγώ είμαι από την κάτω Σαξονία και ξέρω και τη Volkswagen. Και λέτε ότι έχουν εδώ 43 ε, λόμπιστ. Ε, τους εξής τέσσερις βασικά έχουν, οι άλλοι είναι συνεργάτες ε, που ε, ε, ασχολούνται με διάφορα θέματα της εταιρεία. Πρώτον, ξέρετε τη διαφορά ανάμεσα στους λόμπις, στους λόμπις και τους εμπειρογνώμονες που κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Έχετε γνώση αυτής της διαφοράς. Οι πληροφορίες από την Volkswagen είναι αυτές που έγραψαν οι ίδιοι στο Μητρό Διαφάνειας. Δυστυχώς όμως αυτό είναι καθαρά εθελοντικό, δεν παρακολουθείτε πολύ καλά. Ε, βασιζόμαστε λοιπόν στις ίδιες τις επιχειρήσεις ή σε οργανώσεις από τη δική μας ε, να παρέχουν τις ε, σωστές πληροφορίες. Έχουν λοιπόν γράψει εκείνοι 43 ε, λομπίστες ε, και έχουν ε, τέσσερις ε, διαπιστευμένους ε, λομπίστες, αλλά ο λόγος που βρίσκονται εδώ είναι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και με προϋπολογισμό μας τα 3,3 εκατομμύρια. Ε, μα, ακριβώς αυτό είναι το θέμα. Ε, μπορεί να παρεξηγηθεί το θέμα. Σήμερα που ρώτησα ποια είναι η ακρίβεια των φορητών ε, συσκευών, ε, το ποσοστό ανακρίβειας ε, για μένα είναι τεράστιο. Δεν μπορώ να βασιστώ σε αυτά που λέτε εσείς. Γιατί από το 4 στο 43 είναι 90% ποσοστό. Κοιτάξτε, φοβάμαι ότι πρέπει να επαναλάβω αυτά. Δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας. Από το μητρό διαφάνεια τα πήραμε. Σε αυτά βασιζόμαστε. Τι άλλο να κάνουμε. Είναι εθελοντική η εγγραφή. Και ε, στο Μητρό Διαφάνειας ε, ο ορισμός του λόμπι και του λομπίστα είναι αυτούς που προσπαθούν να επηρεάσουν ε, τη νομοθεσία και τη λήψη αποφάσεων. Όταν λέει η ίδια η Volkswagen ότι έχει 43 που κάνουν αυτή τη δουλειά, η ίδια τους χαρακτηρίζει 43. Το γεγονός ότι έχεις ένα μπάζι μια κάρτα για να μπαίνεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν σημαίνει ότι είσαι λόμπι, αλλά ε, συζητήστε το με τη Volkswagen ποιον χαρακτηρίζει η λομπίστα και ποιον όχι από τους υπαλλήλους της. Και αν δεν ισχύει αυτή η πληροφόρηση, ε, ε, αν είναι ανακριβή, σας την αλλάξουν. Εμείς παίρνουμε στοιχεία από το Μητρό Διαφάνεια, σύμφωνα με, τις, με τα ίδια της τα στοιχεία, η ίδια η Volkswagen ε, δηλώνει 43 υπαλλήλους. από το ίδιο το Μητρό διαφάνεια για το πόσοι βρίσκονται τώρα επί τόπου ή δεν βρίσκονται αυτά είναι ε, ε, λεπτομέρειες. Η κυρία Ντελή τελευταία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις σας, η αυτοκινητοβιομηχανία, όπως διαβάζω, το 2014 δαπάνησε πάνω από 18 εκατομμύρια ευρώ. 18 εκατομμύρια ευρώ για λόμπι στις Βρυξέλλες. Η Volkswagen μόνο λέτε έχει 43 λόμπι στις Βρυξέλλες. Πώς είναι απέναντί τους οι ευρωϋπάλληλοι που ε, έχουν ως δουλειά να εφαρμόζουν την νομοθεσία για τις εκπομπές καυσαερίων από τα αυτοκίνητα. Εσείς μπορείτε να το γνωρίζετε να σας πω γιατί τους μέτρησα. Είναι έξι άτομα συγκεκριμένα στο τμήμα αυτοκινητοβιομηχανία και κινητικότητα της Γενική Διεύθυνση Grow που ασχολούνται με τη συγκεκριμένη νομοθεσία για τα μηχανοκίνητα οχήματα και πόσοι στην Αμερική για την προστασία του περιβάλλοντος και του ατμοσφαιρικού αέρα είναι 44. Ιδού λοιπόν το εξή απλό ερώτημά μου. Τι να σου κάνουν έξι άνθρωποι για 500 εκατομμύρια καταναλωτές. Πιστεύετε ότι φτάνουν για την αγορά αυτή. Μήπως για έναν από αυτούς τους λόγους, ή μάλλον είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες που έχουν και υπερβολικό βάρος ως εκπρόσωποι του κλάδου στη λήψη των αποφάσεων. Εντάξει, ε, ε, είναι γεγονό, αλλά λέτε δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπαλλήλου. Εξαρτάται από εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη και πραγματογνωμοσύνη αν δεν έχεις δικού σου εμπειρογνώμονες, τότε εξαρτάται από την αυτοκινητοβιομηχανία και τα κέντρα ελέγχου που χρηματοδοτούνται από την αυτοκινητοβιομηχανία. Αν δεν έχουν δικούς τους εσωτερικούς εμπειρογνώμονες, η αυτοκινητομηχανία αντιστρατεύεται τις μισές προδιαγραφές για τα κόξ και για τα νόξ, το διοξίδιο του άνθρακα και το διοξίδιο ε, του αζότου χρειάζονται ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονε, είναι μακρά πνοή αυτή η διαδικασία. Έχω και άλλη ερώτηση, δεύτερη. Είπατε ότι έγιναν 13 συναντήσεις πέρσι μεταξύ της αρμόδιας Γενική Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Αυτοκινητομηχανίας, χωρίς γραπτά πρακτικά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, κατά την άποψή σα για ποιο λόγο. Πού οφείλεται αυτή η αδιαφάνεια. Γιατί δεν υπάρχουν τέτοια πρακτικά ή δεν είναι προσβάσιμα. Απάντηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κανόνες. Έχουν ένα οδηγό που λέει ότι πρέπει να τηρούνται πρακτικά. Και όταν δεν υπάρχουν πρακτικά ρωτάμε τη Γενική Διεύθυνση Γκρό γιατί δεν εφαρμόζουν το δικό τους κώδικα συμπεριφοράς και δεντολογίας για το πώς ε, συμπεριφέρει στα λόμπι και ποιε είναι οι σχέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι υπάρχουν και κίνδυνοι, βεβαίω, υπάρχουν και ωφέλη από αυτέ τι συναντήσει, ενημέρωση, πραγματογνωμοσύνη. Ρωτήστε τη Γενική Διεύθυνση Grow. Ελπίζω να το κάνετε κιόλα για το πώ εφαρμόζουν του κανόνε αυτού, ποιε είναι οι ασφαλιστικέ ε, δικλείδε και οι διαδικασίε για να εξασφαλίζουν ότι αυτέ οι επαφέ είναι θετικέ και δεν βλάπτουν και δεν καταλήγουν σε αθέμητη επιρροή. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Ολοκληρώνεται η πρωινή συνεδρίαση εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε ε, και με διαφάνεια και με ειλικρίνη απαντήσατε σε αυτά τα θέματα που οδηγούν σε νέα ερωτήματα. Ε, θα τα θέσουμε στους Επιτρόπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν τους δούμε. Το γεγονός ότι υπάρχει υποστελέχωση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Όταν με ρωτάνε όλοι γιατί έχει τρει βοηθού, γιατί του λέω εγώ είμαι καημένη ε, κοινωνιολόγος και έχω ένα σωρό λόμπι από το περιβάλλον μέχρι τη βιομηχανία και αυτό που χρειάζομαι είναι να έχω εμπειρογνώμονες σωστούς ε, ε, εντός της υπηρεσίας μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ραντεβού στι 3 για το δεύτερο μισό ημέρα. Σα Ευχαριστώ πολύ.